Να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση, αν θέλετε. Το πρώτο σημείο είναι η υιοθέτηση της σημερισίας διάταξης. Θέλω να σας ενημερώσω ότι θα αλλάξουμε τη σειρά των σημείων της σημερισίας διάταξης γιατί οι συνάδελφοι ψηφίζουν και σε άλλες επιτροπές ή ψήφισαν σε άλλες επιτροπές. Γι' αυτό αύριο θα αλλάξουμε την έκθεση της ε, Έρικα Μάνερ και του κύριου Μποστινάρου. Πρώτα θα έχουμε την έκθεση Μάνερ και μετά την έκθεση Μποστινάρου. Αν δεν έχετε άλλα σχόλια ή προτάσεις και μετά την ανακοίνωση αυτής της αλλαγής θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε στη μέση διάταξη το χρόνο για κάθε σημείο. Είναι ενδεικτικός αυτός ο χρόνος. Μην θεωρείτε ότι είναι απόλυτος. Μην θεωρείτε ότι κάθε σημείο αρχίζει την ώρα που αναφέρεται ακριβώς, γιατί μπορεί να υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Ούτως ή άλλως δεν ελέγχουμε εμεί πλήρω το χρόνο. Θα ήθελα να πάμε στο δεύτερο σημείο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η εκλογή του τέταρτου αντιπροέδρου της Επιτροπής μας. Ίσως να έχετε ακούσει ο κύριος, ότι ο κύριος Τρεμόπουλος παρετήθηκε από τη θέση του και ο Γενικός Γραμματέας των Πράσινων έστειλε μία επιστολή που προτείνει τον κύριο Νίκο Χρυσόγελο για τη θέση του Αντιπροέδρου. Είναι εδώ ο νέος συνάδελφος, τον καλωσορίζω. Υπάρχουν άλλοι υποψήφοι για αυτή τη θέση. Uh, Άλλη υποψήφια για αυτή τη θέση του τέταρτου αντιπροέδρου. Έχουμε λάβει και τη δήλωση του κύριου Χρυσόγελου, τη δήλωση ενδιαφέροντος. Δέχεστε να είστε υποψήφιος για αυτή τη θέση. Yes, I accept and I would like to thank you. Ευχαριστώ, δέχομαι. Και σας... Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μην προτρέχουμε. θα ήθελα να το κάνουμε διαβοή. Αν υπάρχει ένα υποψήφιο, δεν το κάνουμε διαφορετικά. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση λοιπόν σε αυτή την υποψηφιότητα, θα ήθελα διαβοή να δεχτούμε την υποψηφιότητα του κ. Χρυσόγελου. Μάλιστα, σα εκλέξαμε. Συγχαρητήρια. Δεν έχουμε πολλούς αντιπροέδρους παρόντες σήμερα. Παρακαλώ, ελάτε στο Προεδρείο. Πάμε στο σημείο 3 της τη διάταξης που είναι η έγκριση των πρακτικών της 19 9η, 20 η Δεκεμβρίου και 25 η και 26ης Ιανουαρίου. Ε, Ω έχετε τα πρακτικά. Θα υιοθετηθούν στο τέλος της συνεδρίασης, αν κατά τη διάρκεια της ε, συνεδρίασης δεν υπάρξει αντίρρηση. Πάμε στι ανακοινώσει της Προέδρου. Δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση. Και μπορούμε να περάσουμε πάρα αυτά στο σημείο 5. Έχουμε τη μελέτη της κυρίας Ζουλή Πελεγκράν. I'm να βρω το όνομα του κέντρου αυτού, ε, κέντρο μελετών στο Μιλάνο. Το θέμα της μελέτης είναι προς ένα σύστημα παραχών της πολιτικής για τη συνοχή που να βασίζεται περισσότερο στα αποτελέσματα και τις επιδόσεις. Η κυρία Πελεγκρά. Είναι το κέντρο βιομηχανικών μελετών αυτό στο Μιλάνο. Ε, εγώ ήμουν συντονίστρια της μελέτης αυτής. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ποιο είναι το πλαίσιο. Θα ήθελα να τονίσω ότι η φιλοδοξία της πολιτικής συνοχής είναι να βασίζεται περισσότερο σε επιδόσεις. Και αυτή είναι η βασική συζήτηση που γίνεται τώρα ε, για το μέλλον της πολιτικής αυτής. Δεν είναι νέο επιχείρημα αυτό, αλλά απλώς θα πρέπει να τεθεί στο ευρύτερο πλαίσιο των ε, πολιτικών. Υπάρχουν κάποιες μέθοδοι και κάποιες πρακτικές ε, που προωθούν τη δημόσια διαχείριση που να βασίζεται περισσότερο στις ε, επιδόσεις και στα αποτελέσματα. Ο βασικός στόχος της μελέτης μας είναι να αναλύσει την ε, λογική, τα χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένα σύστημα ή μια πολιτική συνοχή θα βασίζεται περισσότερο στις επιδόσεις και στα αποτελέσματα. Και θα χρησιμοποιεί κάποιους δείκτες και κάποιους μηχανισμούς κινήτρων Πώς μπορεί αυτό να σχεδιαστεί και πώς μπορεί αυτό να εφαρμοστεί. Αυτό είναι το θέμα μας. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω σύντομα τα ερωτήματα της έρευνας και το αναλυτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινηθήκαμε. Είχαμε τρία βασικά ερωτήματα, δύο δέσμες ερωτημάτων που αφορούσαν το σχεδιασμό μιας τέτοια πολιτική που να βασίζεται περισσότερο στα αποτελέσματα, ε, με δείκτες επιδόσεων και μηχανισμούς κινήτρων ενώ η τρίτη δέσμη ερωτήσεων αφορούσε περισσότερο τη διαδικασία καθορισμού μια τέτοια πολιτική, πιο εστιασμένη, πιο προσανατολισμένη ε, στα αποτελέσματα και στι επιδόσει. Λοιπόν, για να χειριστούμε αυτές τις ε, ερωτήσεις, είχαμε ένα αναλυτικό πλαίσιο με τα διάφορα βήματα του κύκλου διαχείρισης των προγραμμάτων. Δηλαδή, ο καθορισμός των στόχων, των δικτών, ο καθορισμός στόχων, παρακολούθηση ε, και μηχανισμοί κινήτρων. Οργανωθήκαμε λοιπόν με βάση αυτόν τον κύκλο των προγραμμάτων ή των σχεδίων. Η μεθοδολογία βασίζεται σε δύο βασικές προσεγγίσεις. Καταρχάς μία ε, μελέτη εγγράφων ξεκινήσαμε ερευνώντας ένα θεωρητικό ολιστικό μοντέλο βασιστήκαμε στο, σύστημα εντολέα εντολοδόχου κάναμε μια πλήρη αναθεώρηση της βιβλιογραφίας και τέσσερις περιπτωσιολογικές μελέτες τέτοιων πολιτικών που είναι εστιασμένες, προσανατολισμένες στα αποτελέσματα και που λειτουργούν αυτή τη στιγμή και που υπάρχουν σε διάφορα επίπεδα, εθνικά, υπερεθνικά ή υποεθνικά. Καταρχάς της Παγκόσμιας Τράπεζας. περίπτωση αυτή έχουμε δύο ε, προγράμματα που εφαρμόζονται αυτή την περίοδο. Ε, ένα πρόγραμμα στην Πολωνία, ένα στην Ιταλία και κοιτάξαμε επίσης και το μοντέλο πολιτικής ανάπτυξης της υπαίθρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η καρδιά της μεθοδολογίας μας βασίζεται σε πολλές συνεντεύξεις που κάναμε με ενδιαφερομένους, με φορείς, ιδίως σε περιφερειακό επίπεδο. Πάνω από 100 συνεντεύξεις κάναμε, 46 με περιφερειακές διοικήσεις, 23 συγγνώμη, και με διάμεσου φορεί 8. Σε εθνικό επίπεδο είχαμε 22 και σε ευρωπαϊκό επίπεδο 7. Επίσης, ε, λάβαμε υπόψη μας και τις απόψεις των ε, ενδιαφερομένων, των δικαιούχων, αν θέλετε, ούτως ώστε ε, να υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Πιστεύουμε ότι η προστιθέμενη αξία της μελέτης μας είναι να καταλάβει το Κοινοβούλιο ποιες είναι οι απόψεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Θεωρούμε βεβαίω ότι γνωρίζετε πολύ καλύτερα τι απόψει των υπαλλήλων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα συμπεράσματα και συστάσει ε, εκπονήθηκαν ε, μετά από το. Μετά από την ε, εξέταση των μελετών, των μελετών και των τεχνικών δυνατοτήτων και κοιτάξαμε επίση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Αυτό το σύστημα εντολέα εντολοδόχου, τι χαρακτηριστικά είχε, πώς το προσεγγίσαμε. Το μοντέλο λέει ότι ένα σύστημα δικτών επιδόσεων ε, είναι πολύ χρήσιμο σε ένα πολυεπίπεδο κυβερνητικό πλαίσιο. Ποιο είναι το επιχείρημα. Ότι οι πληροφορίες ε, δίδονται ασύμετρα σε διάφορα επίπεδα κυβερνητικά στην πολιτική συνοχή. Και έτσι καθίσατε δύσκολο ή αδύνατο να βασιστούμε στην παραδοσιακή αλυσίδα ε, διαβίβασης της εντολής από πάνω προς τα κάτω. Υπάρχουν συμβάσεις όπου οι επιδόσεις των τοπικών φορέων ε, αξιολογείται μέσω δικτών ε, επιδόσεων και μέσω κινήτρων. Τα κίνητρα είναι χρήσιμα ούτως ώστε οι φορείς αυτοί να κάνουν την μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια. Τι μας λέει η θεωρία λοιπόν. Μας λέει ότι πρέπει να υπάρχουν τέτοιοι δείχτες επιδόσεων και ότι πρέπει να υπάρχουν κίνητρα ούτως ώστε να πιέσουμε και να αναγκάσουμε τους φορείς αυτούς σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο να κάνουν μεγαλύτερη προσπάθεια. Ε, πρέπει όμως να υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις για να γίνει κάτι τέτοιο. Πρέπει να υπάρχει, υπάρχει μάλλον αιτιακή σχέση ανάμεσα στην προσπάθεια που κάνει ο τοπικός φορέας και το αποτέλεσμα που πετυχαίνει. Ανάμεσα στην προσπάθεια λοιπόν και στην ανταμοιβή υπάρχει μια σχέση αιτίου αιτιατού. Όταν βλέπουμε τα πρακτικά παραδείγματα το μοντέλο δεν είναι τόσο προβλέψιμο. Από τη μελέτη που κάναμε και από τις ε, περιπτωσιολογικές μελέτες προκύπτει ότι παρότι προσπαθούμε να εφαρμόσουμε ένα σύστημα ε, δικτών επιδόσεων. Η επιτυχία του μηχανισμού κινήτρων ε, δεν είναι δεδομένη. Είναι σπάνια μάλιστα. μάλιστα. Και μάλιστα όπου έχουμε επιτυχία εξαρτάται πάρα πολύ επιτυχία αυτή από το πλαίσιο. Και υπάρχουν κάποιες διευθετήσεις σου εγκαίνερης, ούτως ώστε πραγματικά να έχουμε αυτή την επιτυχία. Αυτό το αποδεικνύω μέσω δύο περιπτωσιολογικών μελετών που είναι πολύ σημαντικές. Δεν θα μιλήσω για την Παγκόσμια Τράπεζα που εδώ στην παρουσίασή μου που βασίζεται περί, περισσότερο σε προϋποθέσεις εξάντε. Δεν ασχοληθήκαμε τόσο πολύ στη μελέτη μας με αυτές. Ε, στην Πολωνία όμως ο μηχανισμός κινήτρων βασίζεται περισσότερο στη συμμόρφωση και στην απορρόφηση των πόρων παρά στα αποτελέσματα. Στην Ιταλία ε, η περίπτωση είναι ενδιαφέρουσα. Στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού έχουν ένα εθνικό σύστημα α, δικτών ε, στις περιφέρειες που καθυστερούν. Υπάρχουν τέσσερις στόχοι ανάλογα με την ε, ποιότητα των υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος, ε, τα παιδιά, ε, φροντίδα για τα παιδιά, φροντίδα για τους ηλικιωμένους, ε, αποκομιδή σκουπιδιών κτλ. και βλέπουν ε, ποιες περιφέρειες ε, υλοποιούν τους στόχους. Θεωρούμε ότι αυτό το παράδειγμα είναι πετυχημένο. Από την ανάλυση της περίπτωση Ιταλίας προκύπτει ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο παράγοντες επιτυχίας που εξηγούν τα καλά αποτελέσματα του συστήματος. Καταρχάς, ε, μία διαδικασία ε, ενεργού συμμετοχής. Εντοπίζουμε και δείχτες και ε, στόχους σε μια διαδικασία από κάτω προς τα πάνω και αρκετά μακροσκελή που κρατάει περίπου δύο χρόνια, που κράτησε αυτή φορά δύο χρόνια από την αρχή της διαδικασίας. Δεύτερον, αυτό που είναι αποφασιστικό είναι η ευελιξία της αξιολόγησης των στόχων που, που τίθενται. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Υπάρχει ένα περίπλοκο σύστημα. Ένα πρόγραμμα θεωρείται επιτυχές ακόμα και αν οι στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί 100% ακόμα και αν το 60% ας πούμε, των στόχων έχουν υλοποιηθεί, θεωρείται ότι το πρόγραμμα είναι επιτυχές εφόσον υπάρχουν κάποιες άλλες προποθέσει, κάποια άλλη όρη που έχουν εκπληρωθεί. Η δεύτερη περίπτωση είναι ενδιαφέρουσα επίσης. Το σύστημα που έχουν υιοθετήσει στην αναπτυξιακή πολιτική. Δεν χρησιμοποιούν ε, μηχανισμό κινήτρων, αλλά ένα σύστημα δικτών πολύ καλά διαρθρωμένο στα πλαίσια της κοινής του κοινού πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης. Κάθε δείχτης συνδέεται με στόχους. Ε, υπάρχει μια λογική παρέμβαση και κάθε δείχτης συγκρίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με άλλα προγράμματα με τους αντίστοιχους δείχτες άλλων προγραμμάτων. Είναι ικανοποιητική η λύση που εξαρτάται όμως από δύο προϋποθέσεις. Καταρχάς, μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα σύστημα γιατί τα προγράμματα διαρθρώνονται με βάση μια φόρμουλα ε, κοινή και υποχρεωτική και δεύτερον γιατί οι παρεμβάσεις είναι σχετικά απλέ σε σχέση με την περιπλοκότητα της πολιτικής συνοχής και των αντίστοιχων προγραμμάτων τη πολιτική συνοχή. Ε, Τώρα, περνάμε στα αποτελέσματα των ημιδιαρθρωμένων συνεντεύξεων, τις ε, οποίες διενεργήσαμε σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Σας παρουσιάζω τα πορίσματά μας για τα διάφορα βήματα του κύκλου διαχείρισης και προγραμματισμού. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις. Ε, το συμπέρασμα είναι ότι η γενική αρχή του να εστιαστούμε στις επιδόσεις ε, είναι γενικώς αποδεκτή από τους εμπλεκόμενους και ότι ένα τέτοιο σύστημα παροχών της πολιτικής συνοχής ε, ε, γίνεται δεκτό. Όμως, Έχουμε διάφορες αντιλήψεις για, τους, για τον όρο της απόδοσης. Ορισμένοι τον θεωρούν ότι αντικατοπτρίζει συμ, ε, ε, συμμόρφωση με συγκεκριμένους οικονομικούς στόχους. Ε, κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι αυτός ο, ο είναι πιο ευρύς και καλύπτει όχι, όχι μόνο ποσοτικά αποτελέσματα αλλά και ποιοτικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, επίδοση είναι η δυνατότητα του προγράμματος να επηρεάσει τους μακροοικονομικούς όρους. Σε ό,τι αφορά τους ε, στόχους και τους δείκτες. Κατά βάση όλοι οι εμπλεκόμενοι ζητούν απλοποίηση της ιεραρχίας ε, των στόχων με λιγότερους και πιο σαφείς στόχους που θα προηγήσουν μετά από διαβούλευση. Επίσης, ε, τα, σύστημα, τα συστήματα δικτών θα πρέπει να απλοποιηθούν με ε, απλούς, λίγους και αξιόπιστους, κυρίως όμως λίγους δείκτες, ε, οι οποίοι να είναι αποδεκτοί από τους εμπλεκόμενους. Πολύ συχνά οι δείκτες αποτελούν ένα περίπλοκο κατάλογο χωρίς πολύ νόημα για τους χρήστες. Τέλος, επικρατεί μια σύγχυση ό,τι αφορά τους τύπους των δικτών και το νόημά τους η διάκριση ανάμεσα σε δείκτες ε, εισόδων, εξόδων, αποτελέσματος και αντικτύπου δεν είναι σαφής σε όλους τους εμπλεκόμενους. Σε ό,τι αφορά την ε, επιλογή, ε, σίγουρα όλοι συμφωνούν ότι η διαδικασία είναι πολύ λεπτής φύσης, αλλά δεν υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα ούτε υπέρ ενός μια συγκρίσιμης υποχρεωτικής λίστας δικτών, ούτε υπέρ μιας ειδική λίστας. Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο τοπικό και το προσφυγικό επίπεδο σε αυτό το θέμα. Σε ό,τι αφορά τώρα τους ε, ε, στόχους, η πιο σημαντική δυσκολία είναι να είναι ρεαλιστική αυτή η στόχη. Οι λύσεις που προτείνονται για το να είναι ρεαλιστικοί στόχη είναι να χρησιμοποιηθούν μελέτες πλαισίου ε, και τεχνικές ε, συμμετοχής, στρογγυλές τράπεζες και διαβούλευση έτσι ώστε να καθοριστούν οι στόχοι στα κατάλληλα επίπεδα κάθε φορά. Σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, η μέτρηση της επίδοσης είναι δύσκολο έργο μέτρηση των επιδόσεων είναι δύσκολο έργο. Το, ε, το σίγουρο είναι ότι η ποσοτική αξιολόγηση και η παρακολούθηση έχουν λάβει ε, μεγάλη προσοχή στο παρελθόν. Ε, δηλαδή, έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε συστήματα δικτών και όχι τόσο πολύ σε συστήματα αξιολόγησης. Οι ποσοτικές μετρήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν με ποιοτικά κριτήρια. Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα των συνεντεύξεων. Και είναι σημαντικό να συνδυαστεί η επαργούση με την αξιολόγηση. Σε εθνικό επίπεδο μας ελέγχθη ότι η αξιολόγηση είναι χρήσιμη όχι μόνο για την, αξιολόγηση, για την μέτρηση επίδοσης, αλλά και για, την, για τον εξυγχρονισμό, για την ενεργοποίηση της αλλαγής. Δηλαδή η αξιολόγηση μπορεί να δώσει και άλλου τύπου φιλοδοξίες, να δημιουργήσει φιλοδοξίες. Επίσης μας ελέγχθη ότι είναι σημαντικό να δούμε το, το χρονισμό και τις πρακτικές λεπτομέρειες, γιατί υπάρχει κάποια δυσφορία σε ό,τι αφορά ε, την εκ αξιολόγηση και το πώς γίνεται. Πολύ συχνά είναι καθυστερεί τόσο πολύ που δεν είναι χρήσιμη για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Επίσης υπογραμμίστηκε η, πολλές φορές η ανάγκη για την ύπαρξη συστημάτων αξιολόγησης που θα είναι ανεξάρτητα και αντικειμενικά. Τέλος, ε, ο κοινός παρανομαστής ήταν ότι ε, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ε, θα πρέπει να, γίνουν, να δημοσιεύονται ευρέως. Σε ό,τι αφορά τους μηχανισμούς κινήτρων. Σε περιφερειακό επίπεδο ε, μας εκφράστηκαν ανησυχίες ότι ε, κάποιοι θα θεωρηθούν υπεύθυνοι ακόμα και για ζητήματα οποία εκφεύγουν της αρμοδιότητάς τους. Οπότε δεν είναι υπέρ ενός συστήματος τέτοιων κινήτρων, ε, ενό δηλαδή αποθεματικού επίδοσης. Κάποιοι άλλοι είπαν ότι τα κίνητρα μπορεί να δημιουργήσουν ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα, δηλαδή οι αρχικοί στόχοι να τίθενται πολύ χαμηλά ε, ή ε, να δίδεται κίνητρο σε πιο συντηρητικές συμπεριφορές για να αποφευθούν οι κυρώσεις. Συνεπώς, αν δοθούν κίνητρα, ε, θα πρέπει να αυτά να λάβουν την μορφή της ανταμοιβή για όποιον εργάζεται καλά και όχι την μορφή Τη ποινή για όποιον δεν εργάζεται σωστά. Για την ακρίβεια προτιμούν οι συντεντευξιαζόμενοι το ένα σύστημα διακύβευση της φήμη περισσότερο και όχι οικονομικά αντικίνητρα. Κίνητρα. Ε, ένα σημαντικό πρόβλημα σε τέτοιου είδους, ε, στην ε, δημιουργία τέτοιων συστημάτων είναι οι υπάρχουσες διοικητικές δυνατότητες. Το, η μείωση του διοικητικού άχθους αποτελεί προτεραιότητα ε, προκειμένου να απελευθερωθούν πόροι και δυναμικό που θα ασχοληθούν με την επίτευξη των αποτελεσμάτων. Ε, πολλοί από όσους μας μίλησαν μας ε, τόνισαν την ανάγκη αλλαγής στην φιλοσοφία της εφαρμογής πολιτικής συνοχής. Λένε ότι ένα σύστημα προσανατολίζεται πιο πολύ στην απόδοση και στα αποτελέσματα θα πρέπει ε, να δίνει περισσότερη σημασία στα ίδια τα αποτελέσματα και λιγότερο στις διαδικασίες. Κάποια άλλα συμπεράσματα είναι τα εξής. Ένα τέτοιο σύστημα δεν μπορεί να ε, είναι μοναδικό και ενιαίο για όλους, ομοιόμορφο. Χρειάζεται να ληφθούν υπόψη τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των διαφορετικών προγραμμάτων και εθνικά χαρακτηριστικά. Για παραδείγμα, ε, διαφορετικές προσεγγίσεις ε, σε ό,τι αφορά την κουλτούρα της κάθε χώρας καθώς επίσης ε, και τα διαφορετι... η διαφορετική διοικητική δομή, αν μια χώρα είναι ομοσπονδιακή ή όχι, η διοικητική δομή, αν είναι πιο αποκεντρωμένη, πιο συγκεντρωτική κλπ. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, έτσι ώστε να μην έχουμε ένα ομοιόμορφο σύστημα ε, παροχών. Εδώ πέρα βλέπετε κάποιες ε, καινοτόμες προτάσεις που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις. Για παράδειγμα, ένα πρωτόκολλο παρακολούθησης της, ε, των επιδόσεων που θα περιλαμβάνει διάφορες λεπτομέρειες για το σύστημα παρακολούθησης. Για παράδειγμα, η φύση των στόχων, αν μπορούν να αναθεωρηθούν ή όχι κλπ. Τέτοιου είδους χαρακτηριστικά. Επίσης, η χρήση επίσημων στατιστικών πηγών προτάθηκε πολλές φορές αντί να βασιζόμαστε μόνο στην παρακολούθηση και τα δεδομένα προκύπτουν από αυτήν. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση από την άλλη μεριά έγινε η πρόταση να διεξάγεται η αξιολόγηση τουλάχιστον δύο-τρεις φορές σε τακτικά στάδια κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και της υλοποίησης του προγράμματος. για παράδειγμα στο 30% της υλοποίησης, στο 40% και μετά στο 70%. Και τέλος βέβαια όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Έχετε πιο πολλές λεπτομέρειες πάνω στις διαφάνειες, δεν θα επισέλθω σε αυτό. Νομίζω ότι προχώρησα πολύ γρήγορα. Ωραία, συμπεράσματα της μελέτης. Ε, καταλήξαμε στο ότι ε, η θέσπιση ενός ε, συστήματος, τέτοιου συστήματος παροχών απαιτεί να αλλάξουμε την εστίαση από την συμμόρφωση και τις δαπάνες και να, την, ε, και να εστιαστούμε πιο πολύ στα, στις και τα αποτελέσματα. Αυτό έχει υπέρ και κατά. Χρειάζεται μια ε, ριζική αλλαγή στην ε, διοικητική νοοτροπία πριν μπούμε σε τεχνικά ζητήματα για το ποιους δείκτες θα επιλέξουμε, πώς θα τους επιλέξουμε, ε, αν οι στόχοι θα είναι αναθεωρήσιμοι ή όχι κλπ. Χρειάζεται μια αλλαγή στη φιλοσοφία και στην οτροπία. Μια λύση είναι να ενεργοποιήσουμε σε τοπικό, περιφερειακό, και εθνικό επίπεδο την πολιτική σφαίρα, τους πολιτικούς. Χρειάζεται επίσης μια συνολική προσέγγιση που δεν θα βασίζεται μόνο σε μετρήσεις επιδόσεων ένα τέτοιο σύστημα παροχών που θα εστιάζεται στις, ε, στα αποτελέσματα είναι ένα πακέτο κατά βάση που περιλαμβάνει όλες τις διαφορετικές φάσεις ε, του κύκλου διαχείρισης του προγράμματος από την επιλογή των προγραμμάτων στον εντοπισμό των στόχων κλπ. Οι επιδόσεις δεν θα πρέπει απλώς να αξιολογούνται αλλά και να δημιουργούνται μας είπε κάποιος από αυτούς που μας έδωσαν συνέντευξη. Θα πρέπει λοιπόν να βλέπουμε όλες τις διαφορετικές φάσεις και να εφαρμόσει αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ευελιξίας, της συμμετοχής και της ίδιας ευθύνης σε όλες αυτές τις φάσεις. Άλλο συμπέρασμα είναι ότι μια ισορροπημένη προσέγγιση θα πρέπει να ε, συνδυάζει τους δείκτες με την αξιολόγηση. Δεν είναι το ένα εις βάρος του άλλου η απλοποίηση του λογικού πλαισίου της ε, πολιτικής ε, συνοχής και του συστήματος παραχών της πολιτικής συνοχής είναι απόλυτα απαραίτητη. Ε, θα πρέπει το σύστημα παροχών να συνδυαστεί με το επίπεδο προγραμματισμού. Γιατί αυτό έχει σχέση με την, το, τη σχέση δικτύου αιτιατού ε, η οποία είναι πιο εύκολα να προσδιοριστεί σε επίπεδο προγράμματος. Εκεί το κατάλληλο σημείο στο οποίο θα εφαρμόσουμε αυτό το σύστημα παροχών. Άλλο συμπέρασμα, δείκτες αποτελέσματος ε, θα είναι η πιο κατάλληλοι για ένα τέτοιο είδου σύστημα που θα βασίζεται στα αποτελέσματα και τις επιδόσεις. γιατί πραγματικά αυτοί οι δείκτες αποδεικνύουν και αντικατοπτρίζουν ε, την επιτυχία των ε, πολιτικών και των στόχων. Ε, σε ό,τι αφορά το σύστημα κινήτρων, είναι δύσκολο να εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως, όπως θα δείτε και στην επόμενη διαφάνεια, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με την εφαρμογή εθελοντικής ε, φύσεως αποθέματος ε, ε, για τη για, που, θα δίδεται σε αυτούς που έχουν παρουσιάσει καλύτερες επιδόσεις ε, υπό βέβαια συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις Ε, θα μπορούσαμε να επιβάλλουμε θα μπορούσαν να επιβληθούν κυρώσει αν τα κράτη-μέλη ε, δεν σέβονται και δεν συμμορφώνονται με το πλαίσιο επιδόσεων. Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί, ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε χώρας σε επίπεδο προγράμματος. Επί αυτής της βάσης έχουμε ε, υποβάλει και κάποιες συστάσεις. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να βασιστούμε σε δύο σκέλη. Πρώτον, το πολιτικό σκέλος, όπου χρειάζεται ε, να προωθήσουμε μια, ένα πραγματικό διάλογο, πολιτικό στατικό διάλογο για την ε, πολιτική συνοχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για παράδειγμα, με τη δημιουργία ενός Συμβουλίου Συνοχής όπως το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης θα πρέπει να δώσει περισσότερη ε, σημασία στα, σε επιδόσεις και στα αποτελέσματα. Δεύτερο σκέλος, το διοικητικό σκέλος. Χρειάζεται να μειώσουμε ε, τα κριτήρια ε, συμμόρφωσης και ε, να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες. Εδώ, εδώ μπορεί να γίνει μια ένα πραγματικά καινούριο συμβόλαιο New Deal. Ε, ένα πραγματικό σύστημα μέτρησης και αξιολόγησης σε επίπεδο προγράμματος με ποσοτικές αξιολογήσεις της προόδου του προγράμματος βασισμένες σε τρεις κατηγορίες δικτών input, output και αποτέλεσμα και δεύτερον αξιολόγηση των επιδόσεων του προγράμματος σε ό,τι αφορά ε, την, με την ενεργοποίηση διαφόρων δραστηριοτήτων αξιολόγησης δεν θα εμπλέκαμε το ε, επίπεδο του project ε, μόνο εθελοντικά και τρίτον θα συστήναμε να υιοθετηθεί ένα σύστημα προϋποθέσεων σύμφωνα με το οποίο η πρόσβαση στη χρηματοδότηση θα συναρτάται από την καθιέρωση ενός πλαισίου αξιολόγησης και παρακολούθησης όπως αυτό που ανέφερα προηγουμένως για να λειτουργήσουν αυτές οι συστήσεις χρειάζονται κάποια, να ληφθούν κάποια, χρειάζεται να ληφθούν κάποια μέτρα τα οποία είναι πραγματικά χρήσιμα ε, και απαραίτητα. Θα σα αναφέρω ποια είναι αυτά. Πρώτον, επικοινωνία και διαφάνεια. Το αποτελέσματα των αξιολογήσεων θα πρέπει ε, να δημοσιοποιούνται και να διαδίδονται. Και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και στον πολιτικό διάλογο. Για παράδειγμα, μια πλατφόρμα στο ίντερνετ η οποία θα δημοσιοποιεί ακριβώς αυτά τα στοιχεία θα μπορούσε ε, ε, να είναι πολύ χρήσιμη με μετάφραση στα αγγλικά των το, το, συνόψεων. Επίσης, ε, ένα σύστημα το οποίο θα εστιάζεται πιο πολύ στην απόδοση. Αυτό έχει επιπτώσεις ό,τι αφορά τον προπολογισμό. Και θα πρέπει να φύγουμε από την αξιολόγηση της συμμόρφωσης για να κοιτάξουμε τι γίνεται σε άλλο επίπεδο. Αυτό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Επίσης, έχει νομικές επιπτώσεις. Η αρχή αυτή θα πρέπει νομικά να κατοχυρώνεται στην καινούργια κανονισμό και στους καινούργιους κανονισμούς για την ε, περιφερειακή συνοχή. Επίσης, κάθε πρόγραμμα θα πρέπει να εστιάζεται σε περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων δένοντας αν θέλετε και το σύστημα των δικτών όλα αυτά σε ένα, με έναν τρόπο που θα εμπλέκει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς όχι μόνο για να τεθούν οι σωστοί δείκτες αλλά και για να αποκαλύπτονται σωστά οι προτιμήσεις. Επίσης η αναθεώρηση από τους ομοτήμους αποτελεί επίσης μια αρχή που θα πρέπει να γίνει σεβαστή η ανεξαρτησία και η αξιοπιστία θα πρέπει να διασφαλίζονται, για παράδειγμα μέσω της ίδρυσης ενός εθνικού σώματος που θα ε, είναι αρμόδιο σε τέτοιο επίπεδο προγραμματικό και το κριτήριο της ποιότητας ε, των σωμάτων αυτών θα πρέπει να ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο ρόλος τώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να παρέχει ε, καθοδήγηση για τα πρότυπα και τις μεθοδολογίες ποιότητας και να διασφαλίζει ότι κινητοποιείται επαρκής ε, διοικητική ικανότητα στα κράτη-μέλη. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις οι τοπική και εθνικοί εμπλεκόμενοι φορείς μας αναφέρουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ρόλο καθοδήγησης για στρατηγικά θέματα και υποστηρικτικό ρόλο σε καινοτομικά θέματα, το οποίο και φθήνει τον τελευταίο καιρό. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα, όπως ανέφερα, θα πρέπει να επικεντρωθεί στα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται παρά σε θέματα συμμόρφωσης και προς το σκοπό αυτό θα μπορούσε να ιδρύσει τακτικά φόρουμ για συζήτηση των αποτελεσμάτων, για παράδειγμα της Επιτροπής Ρέτζη, ειδικά για τέτοια θέματα ή ένα, μια συνάντηση κάθε δύο χρόνια και πάλι ίσως μια συνάντηση με την Επιτροπή των Περιφερειών θα πρέπει να χρησιμοποιεί πιο συστηματικά και τακτικά τέτοια τα αποτελέσματα να συμβάλλει σε μια online πλατφόρμα όπως ανέφερα και να χρησιμοποιήσει το ρόλο του ως συνομοθέτης για να διασφαλίσει ότι οι καινοτομίες ε, ε, περιλαμβάνονται σε όλους τους κανονισμούς μετά το 2013 τώρα για τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν και αυτό το ρόλο τους, ιδιαίτερα η την των Περιφερειών. Θα πρέπει να δώσουν μια πλατφόρμα για τη συζήτηση και τη ε, συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων. Συγγνώμη, ξέχασα να σας πάω στην ε, κατάλληλη διαφάνεια. Βλέπετε τώρα σε ένα πίνακα το διάφορο σενάρια που προτείνει η μελέτη και έχω τονίσει κάποια θέματα σε ό,τι αφορά τους στόχους, την επικέντρωση σε περιορισμένους στόχους, σε ό,τι αφορά τις ε, δείκτες, ε, output ε, και οι σχετικοί δείκτες, λίγοι δείκτες σε επίπεδο προγραμματικό. Κάποιοι δείκτε για τα αποτελέσματα μπορεί να είναι κοινοί για όλα τα προγράμματα, κάποιοι άλλοι θα πρέπει να είναι συγκεκριμένοι ανάλογα με το πρόγραμμα. Τώρα για του στόχου θα πρέπει να είναι αναθεωρήσιμοι. Θα πρέπει να καθορίζονται με συμμετοχική διαδικασία και η χρήση στατιστικών στοιχείων είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ενθαρρυνθεί. Δεχτήκαμε την ιδέα δημιουργίας ενός πρωτοκόλου αξιολόγησης της απόδοσης για, για να βελτιωθεί η δέσμευση των εμπλεκομένων φορέων. Επίσης θεωρούμε ότι ένα εθνικό σώμα το οποίο θα εξασφαλίζει θέματα ανεξαρτησίας θα πρέπει να συσταθεί σε ό,τι αφορά τους μηχανισμούς κινήτρων τώρα. Συστήνουμε τη ίδρυση ενός υποχρεωτικού συστήματος ερεσιμότητας, δηλαδή τα κράτη-μέλη που δεν θα ακολουθούν τις συστάσεις για ένα πλαίσιο αξιολόγησης, δεν θα έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Αλλά δεν συστήνουμε τη δημιουργία δεσμευτικών αποτελεσμάτων. Νομίζω ότι ως επιλογή θα μπορούσε αυτό να εφαρμοστεί σε προγραμματικό επίπεδο εφόσον υπάρχουν και συντρέχουν οι λόγοι. Και τώρα να συγκρίνω το σενάριο αυτό με την τρέχουσα πρόταση που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σχετικό κανονισμό που δημοσιεύθηκε το φθινόπωρο. Υπάρχουν πολλά κοινά σημεία. Για παράδειγμα, η ανάγκη εστίαση σε περιορισμένο ρυθμό καλά ορισμένων στόχων, ε, ο ορισμός των δικτών, input-output, αποτελέσματα, η χρήση δεστικών στοιχείων, ε, συμμετοχική μέθοδος. Κάτι άλλο κοινό είναι η πρόταση να καταστεί δεσμευτική η έγκριση της σχετικού πλαισίου να τεθεί η Υπάρχουν διάφορα στοιχεία τα οποία δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ασύμβατα με το δικό μας σύστημα, για παράδειγμα η μακροοικονομική ρεσιμότητα. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες σημαντικές διαφορές. Η πιο σημαντική εξ αυτών έχει να κάνει με την πρόταση της ε, ε, Επιτροπής να δημιουργηθεί ένα αποθεματικό υποχρεωτικό 5% σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση για τα κράτη-μέλη. Η πρόταση αυτή περιλαμβάνεται στο άρθρο 18, 19 και 20 του σχετικού κανονισμού. Αυτή είναι η πιο βασική διαφορά. Υπάρχουν και άλλες διαφορές οι οποίες είναι πιο βαθμιαίες αν θέλετε έχουν να κάνουν πιο πολύ με θέματα έμφασης, παρόλα αυτά είναι σημαντικές όμως. Για παράδειγμα, η μελέτη αυτή επιμένει στο ευρύτερο πλαίσιο πολιτισμικής αλλαγής που χρειάζεται για να υπάρχει ένα σύστημα που θα εστιάζεται πιο πολύ στα αποτελέσματα. Ζητά μετατόπιση από τη συμμόρφωση προς τη συμμόρφωση και όντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλει πολλές προσπάθειες προς την κατεύθυνση της απλούστευσης, της απλοποίησης, αλλά ίσως δεν έχει τονίσει αρκετά την πολιτική συνάφεια, την πολιτική σημασία των αλλαγών αυτών, των προτινόμενων αυτών αλλαγών. Άλλες διαφορές τώρα σε ό,τι αφορά θέματα έμφασης. Η μελέτη επιμένει σε θέματα ε, διάδοση των αποτελεσμάτων και των πολιτικών τους συνεπειών. Θεωρούμε ότι αυτή η πολιτισμική, αν μετατόπιση, αλλαγή που σας ανέφερα, θα είναι επιτυχής αν η πολιτική σφαίρα έχει πρόσβαση σε ό,τι αφορά τη χρήση των αποτελεσμάτων αυτών της αξιολόγησης. Ευχαριστώ. Thank you. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για τις συστάσεις ε, που μας αναφέρετε και για το γεγονός ότι εξετάσατε και την τρέχουσα πρόταση. Να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, αν έχουν οι συνάδελφοι ερωτήσεις, απορίες. Έχουμε μαζί μας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιτροπή. Θα ήθελα να σας δώσω το λόγο μετά να πείτε δύο λόγια, αλλά να ξεκινήσουμε με μία ερώτηση ίσως, επειδή αναφέρετε, το είπατε κιόλα, ότι θα πρέπει να γίνει μια μετατόπιση, να κοιτάξουμε πέρα από το σύστημα ε, συμμόρφωσης με τους κανόνες. Να μετατοπιθούμε λοιπόν από τα κριτήρια απορρόφησης σε μια προσέγγιση βασισμένη στα αποτελέσματα. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον ασφαλώς, αλλά δεν μπορούμε να το πληρώσουμε απαραίτητα. Θα πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία λοιπόν μεταξύ της σημασίας της ε, της συμμόρφωσης, της απορρόφησης και των αποτελεσμάτων μιας πολιτικής. Αυτή είναι μια αμφιβολία που έχω σε ό,τι αφορά τα όσα μας παρουσιάσατε. Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει και αυτό με το γεγονός ότι προκειμένου να υπάρχει μια προσέγγιση βάση αποτελεσμάτων, Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε τον τρόπο που αξιολογούνται οι πολιτικές από όλα τα θεσμικά όργανα και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξετάσει άλλες πτυχές και καθαρά την ε, πτυχή της χρηματοδότησης σε ό,τι αφορά την ε, απορρόπηση των ε, διαθέσιμων κονδυλίων. Επίσης θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να δικαιολογηθεί και η μετατόπιση σε εθνικό επίπεδο, να μην υπάρχει πολιτικό και οικονομικό κόστος σε ό,τι αφορά τη διαφορά αυτή στην απορρόφηση. Θα πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν και πέρα από το σύστημα τι γίνεται και πέρα από το σύστημα να κινηθούμε προς μία πολιτική βάση των αποτελεσμάτων. Θα ήθελα να ακούσω και τα σχόλια τα δικά σας από αυτό. Το δεύτερο θέμα, σε σχέση με αυτά που μας αναφέρατε, είπατε ότι έχουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τον κατάλογο των δικτών. Και στις συζητήσεις που είχαμε, εκφράστηκαν πολλές αμφιβολίες σε ό,τι αφορά την γενική φύση των δικτών που προτείνονται για την επόμενη αυτή περίοδο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίθηκε, αντέδρασε σε αυτές τις αμφιβολίες ως εξής. Χρειαζόμαστε την ικανότητα για να ομαδοποιούμε και για να συγκρίνουμε και αν έχουμε πολύ συγκεκριμένους δείκτες ε, για πολύ μικρά προγράμματα, για πολύ μικρές περιφέρειες θα χρειαζόμαστε και συγκεκριμένους ε, δείκτες. Αλλά πώς είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η ομαδοποίηση. Αυτή λοιπόν η αντίθεση αποτελεί ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να δούμε πώς θα επιλύσουμε. Αν θέλετε να σχολιάσετε. Και κατά τρίτον, όλοι συχνά λέμε ότι αν ε, οριστούν οι δείκτες αυτοί για να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα, οι φιλοδοξίες θα είναι πολύ χαμηλές. Πώς μπορούμε λοιπόν να διαφύγουμε από αυτό το δίλημα. Αν θα θέλετε να σχολιάσετε λοιπόν. Και συνάδελφοι, όποιος θέλει να πάρει το λόγο. Αν δεν θέλετε το λόγο, να πάρει το λόγο. Α, μάλιστα, ο κύριος, ε, ο Βίκτορ έχει το λόγο. Ε, some comments. First, I would... Ε, Κάποια σχόλια. Καταρχάς, Νόμιζα ότι η μελέτη σας θα τονίσει και την ανάγκη βελτίωσης των θεσμικών και αντικειτικών ικανοτήτων, γιατί προτού ζητηθεί οποιαδήποτε περαιτέρω βελτίωση της ικανότητας, της ικανότητας για καλύτερο σχεδιασμό των project, θα πρέπει να κοιτάξουμε τι γίνεται και στο ιστορικό των εθνικών κρατών μελών, των περιφερειών, όπου συχνά δεν υπάρχει η απαραίτητη διοικητική ικανότητα για τον σχεδιασμό των έργων. Στην μελέτη αυτή δεν υπάρχει αναφορά οποιαδήποτε τέτοια της δραματικής αυτής ανάγκης και αυτό μάλιστα για την περίοδο πριν το 2014. και το 2014 θα εφαρμοστεί όλος ο μηχανισμός αυτός. Θα βρισκόμαστε σε φάση, αν θέλετε, ε, εφαρμογής των λεπτομεριών Κατά δεύτερον, οι δείκτες που αναφέρατε προηγουμένως, πολύ καλοί, αλλά δεν έχουμε λεπτομέρειες. Πόσο και ποια είναι τα αντικειμενικά κριτήρια για να αποφευχθούν ε, το περιθώριο, αν θέλετε, λιγμών ή υποκειμενικές ερμηνείες, γιατί στην περίπτωση αυτή μπορεί τα κονδύλια αυτά να μεταφέρονται στις Βρυξέλλες χωρίς ε, να υπάρχει σωστός λόγος. Κατά τρίτον, τι θα γίνει με το 5% αποθεματικό απόδοσης, γιατί στην Επιτροπή Ρέτζη Περιφερειακής Ανάπτυξης μας είπαν ότι τα χρήματα αυτά θα παραμείνουν στο ιστορικό των κρατών μελών και αντιθέτω, ο προπολογισμό, η Επιτροπή Προπολογισμών μα διαβεβαίωσε ότι όχι, τα χρήματα αυτού του παθηματικού θα μεταφερθούν στι Βρυξέλλε. Εγώ θεωρώ ότι εδώ θα είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα αυτό και θα υπάρχει σοβαρό καυγά. Αν το αποδεχτούμε αυτό. Και τέλο, ε, το μέθο τη κρίση θα δούμε και μακροοικονομικές, μακροοικονομικούς όρους που συμπίπτουν κατά κάποιον τρόπο με το six-pack και την ε, συνθήκη για την χρηματοοικονομικό συμβόλαιο. Δηλαδή συνεχίζουμε να τιμωρούμε τις περιφερειές. Δεν είναι αυτός ο στόχος της πολιτικής συνοχής και το κοινοβούλιο. Αντίθετο στην ιδέα αυτή. Πέντε σημεία. Όχι μόνο είναι υπερβολικό, αλλά με πολύ ασαφή κριτήριο μάλιστα και με δραστική μείωση του προϋπολογισμού λόγω των του αυτού ορίου μόνο 2,5% αλλά σε εποχές που το ΕΕΠ συρρυκνώνεται ε, ίσως λίγο σε μεγάλα κρατημέλη, ίσως πολύ σε κάποιες φτωχές χώρες. Πιο λίγα χρήματα και πιο πολλές κυρώσεις. Και πάλι αυτό δεν αποτελεί την φιλοσοφία της πολιτικής συνοχής. Πώς θα συμπληρωθούν λοιπόν αυτές οι δύο τάσεις προκειμένου να ωφελήσουν την πολιτική συνοχής που σκοπό έχει να εξαλείψει τις διαφορές και όχι να τις οξύνει όπως γίνεται σήμερα. Ευχαριστώ. Thank you. Um, Ευχαριστώ. Ένα σύντομο σχόλιο. Ανοίγει πολλές συζητήσεις η έκθεση αυτή και αυτό είναι σημαντικό. Όταν λέμε θα εστιάσουμε στα αποτελέσματα. Όλοι συμφωνούμε με αυτή τη λογική. Από τη δική μου εμπειρία, από την σουηδική εμπειρία, ε, τα αποτελέσματα είναι καλύτερα, μπορώ να πω, εάν οι τοπικοί, περιφερειακοί φορείς, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι εταιρείε, όλοι οι ενδιαφερόμενοι εμπλέκονται και στον προγραμματισμό. Κάπου το αναφέρατε αυτό ότι είναι σημαντικό για τα αποτελέσματα, αλλά ε, εν συνεχεία δεν το είδα πιο ανεπτυγμένο. Αν εμπλέξουμε όλους αυτούς τους φορείς στον προγραμματισμό, τα αποτελέσματα είναι καλύτερα. Από τη δική μου εμπειρία αυτό προκύπτει. Συμφωνείτε εσείς με αυτό? Σας ευχαριστώ. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα. Ότι το σύστημα θα πρέπει να εστιαστεί πιο πολύ στα αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι κάποιες από τις συστάσεις κινούνται προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Αφενός, θέλουμε το διοικητικό άχθος να μειωθεί, αλλά αφετέρου γίνεται μία σύσταση αξιολόγησης, δις και τρεις κατά τη διάρκεια ενός project και σύσταση σχετικών εκθέσεων. Όλα αυτά δεν συνάδουν το ένα με το άλλο. Ένα δεύτερο θέμα είναι οι εθνικές αρχές αξιολόγησης. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το α, διευκρινίσουμε, να το περιγράψουμε με λεπτομέρεια και αυτό δεν βλέπω να υπάρχει στην έκθεση. Ένα άλλο θέμα είναι η συζήτηση των αποτελεσμάτων στον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερο στην Επιτροπή των Περιφερειών. Θα ήταν καλό να ενημερώνεται η Επιτροπή των Περιφερειών για τα αποτελέσματα αυτά, αλλά δυσκολεύομαι να, φαντάζω, δυσκολεύομαι να φανταστώ μια κοινή συζήτηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, γιατί πρόκειται για ένα μεγάλο θέμα ε, και θα σήμαινε πάρα πολύ δουλειά. Θα θέλετε να το σχολιάσετε όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ε, Κυρία Πελεγκρέν, έχει το λόγο. Πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία, όντως. μεταξύ αντιτιθέμενων ή συγκρουσιακών δυνάμεων, και είναι η λέξη πολύ ισχυρή. Καταρχάς, να υπάρξει συμμόρφωση με τους κανόνες και συνεχεία να υπάρχουν αποτελέσματα. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πιο τολμηροί και να αναγνωρίσουμε ότι όταν έχουμε δημοσιονομικές, δημοσιονομικούς περιορισμούς, κάποια επιλογή πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Και για να μειώσουμε το διοικητικό άχθος που βαραίνει τις τοπικές αρχές και τους φορείς αυτούς και τους δικαιούχους, Υπάρχουν εργαλεία όπως της αναλογικότητας που το προτείνει, εργαλείο, ε, το προτείνει η Κομισιόν αυτό το εργαλείο. Ή προτείνει να χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένοι κανόνες επιλεξιμότητας. Όντως πρέπει να βρεθεί λοιπόν μια ισορροπία. Δεν θέλουμε να ξεχάσουμε ότι πρέπει να ελέγξουμε πραγματικά την συμμόρφωση, αλλά υπάρχουν κανόνες. Και η Κομισιόν θα πρέπει να έχει περισσότερη εμπιστοσύνη στα κράτη-μέλη ότι λειτουργούν καλά και να απελευθερώσει έτσι πόρους, ούτως ώστε να κινηθούν προς την επίτευξη αποτελεσμάτων. Υπάρχει ένα δίλημα, όπως είπατε, ανάμεσα στα, στις ειδικές ανάγκες και στην, σε κάποιες γενικές προϋποθέσεις που θα ισχύουν για όλα τα προγράμματα, για όλες τις χώρες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η μελέτη μας βασίζεται σε διαβουλεύσεις που είχαμε πολλούς περιφερειακούς και τοπικούς φορείς και αρχές. Και γενικά είδαμε ότι είναι αρκετά απρόθυμοι ε, να συμμορφωθούμε οτιδήποτε ε, επιβεβλημένο, υποχρεωτικό κτλ. Ίσως υπάρχει μια προκατάληψη δηλαδή προς σε αυτό το, αυτήν την κατεύθυνση, αλλά αξίζει τον κόπο να τους ακούσουμε. Το πρόγραμμα θα πρέπει να το δούμε σε ένα πλαίσιο ανάλυσης και δράσης σαν, μια, σαν ένα πακέτο. Αυτή είναι μια λύση, γιατί εκεί ξέρουμε πολύ καλά σε ποιον ανήκει το πρόγραμμα, ποιος κάνει τις παρεμβάσεις και βλέπουμε και αυτά τα αποτελέσματα Υπάρχει παρέμβαση, αποτέλεσμα. Όλοι εξαρτώνται από την εμπλοκή και τη διαβούλευση με τους ε, stakeholders, με τους ενδιαφερόμενους. Και ίσως ε, πρέπει να βασιστούμε στο κάθε πρόγραμμα, δηλαδή σε επίπεδο προγράμματος για να λύσουμε όλα αυτά τα διλήμματα που ακούστηκαν. Uh, uh, Επίσης, μία δέσμη στόχων Μπορεί αυτό να μας παραπλανήσει. Οι στόχοι μπορεί να μας πλανήσουν. Αλλά αν εμπλέξουμε τους ενδιαφερόμενους φορείς, τους stakeholders, στον καθορισμό αυτών των στόχων, πραγματικά μπορούμε να πετύχουμε ε, στόχους που μας ενδιαφέρουν, ε, τίμιους, ε, όχι οπορτουνιστικούς κτλ. Επίσης, η Κομισιόν προτείνουμε να αξιολογήσει το αν υπάρχει το θεσμικό δυναμικό σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό το δυναμικό αυτό. Και φυσικά πρέπει να αξιολογείται για τους δείκτες. Η Κομισιόν πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο εδώ και να δώσει καθοδήγηση, να καθορίσει τη μεθοδολογία Δικός τους είναι αυτός ο ρόλος. Τώρα, για το αποθεματικό που ενεργοποιείται με βάση επιδόσεις. Δεν μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Αυτό είναι η δουλειά της Κομισιόν. Δεν μπαίνω σε αυτά τα χωράφια. Και οι μακροοικονομικές ε, προϋποθέσεις. Ακούω τα επιχειρήματά σας ότι αυτό μπορεί να είναι αρνητικό για τις περιφέρειες. Ε, οι περιφέρειες όμως δεν είναι αυτές που δημιούργησαν την κατάσταση. Αυτό μας θυμίζει το επιχείρημα για το ποιος έχει τις ευθύνες. Εμείς για αυτό το σημείο δεν, δεν ρωτήσαμε τους τοπικούς φορείς. Πάντως πρέπει να υπάρχει λογοδοσία, κατανομή ευθυνών. Δεν ασχολήθηκε όμως η μελέτη με αυτό. Έχουμε καλύτερα αποτελέσματα αν οι τοπικοί φορείς εμπλέκονται στον προγραμματισμό. Καλή ερώτηση. Η πρώτη εύκολη απάντηση είναι ναι, προφανώ χρειαζόμαστε μεγαλύτερη εμπλοκή από πλευρά του. Αυτό είναι κάτι που το λέμε και το ξαναλέμε και το ξαναλέμε προφανώ. Αυτό ισχύει για τον καθορισμό των δικτών και των στόχων. Βέβαια, εδώ πρέπει να δούμε και τι συμφέροντα υπάρχουν. Πρέπει να αξιολογήσουμε, πρέπει να κατευθύνουμε την όλη διαδικασία, ώστε να υπάρχει συνένεση στο τέλος της ε, διαβούλευσης ό,τι αφορά τους στόχους του προγράμματος. Λέει... Ελπίζω να απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Βερόνικα Γκάτι. Ευχαριστώ κυρία Φίμπνερ. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνετε να συμμετάσχουμε και εμείς στη συζήτηση και να απαντήσουμε αλλά κυρίως ευχαριστούμε πολύ για την πρωτοβουλία να παραγγείλετε αυτή τη μελέτη. Νομίζω ότι θα συνεισφέρει πάρα πολύ στην, ε, διαδικασία διαλόγου. Μόλις έλαβα την έκθεση, συνεπώς δεν μπορώ να σχολιάσω λεπτομερώς, αλλά ε, άκουσα την παρουσίασή της ε, και η μελέτη μας βρίσκει σύμφωνους εμάς την Κομισιόν σε πάρα πολλά σημεία, σαν όχι σε όλα. Κοιτώντας τα συμπεράσματα, εστιάζονται σε πολλά σημεία τα οποία συζητούνται και εδώ στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Συνεπώς είναι πραγματικά πολύ χρήσιμη αυτή η μελέτη. Η εστίαση στα αποτελέσματα είναι ένας ε, βασικός άξονας της μεταρρύθμισης. Δεν θα συμφωνήσω πλήρω με αυτό που είπε η Ζουλή, ότι δεν αναγνωρίζουμε την αλλαγή της νοοτροπίας που χρειάζεται, που είναι απαραίτητη. Όχι, την αναγνωρίζουμε. Ε, ίσως δεν βρίσκεται στο ίδιο το κείμενο των ρυθμιστικών προτάσεων, αλλά σίγουρα αναγνωρίζουμε ότι η εστίαση στα αποτελέσματα και τις επιδόσεις χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας. Αυτό που επιζητούμε είναι να περιγράψουμε καλά το ποιοι είναι στόχοι και μετά να παρακολουθήσουμε την πρόοδο. Αυτό αυτή τη στιγμή δεν λαμβάνει χώρα επαρκώς. Γιατί, ακριβώς όπω είπατε, εστιαζόμαστε πιο πολύ στην απορροφητικότητα και τη συμμόρφωση με τους χρηματοοικονομικούς κανονισμούς. Ο κίνδυνος είναι ότι αν συνεχίσουμε μόνο σε αυτό το δρόμο, θα καταλήξουμε να δαπανούμε σωστά του πόρου μα αλλά χωρίς να επιτυγχάνουμε επαρκές αποτέλεσμα. Και βέβαια αυτό δεν είναι το επιθυμητό σε ένα περιβάλλον περικοπών και περιορισμένου προϋπολογισμού. Πληροφοριακά επίσης να σας πω ότι η DG Regio έχει ξεκινήσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα για την δοκιμή του συστήματος εστίασης ε, σε αποτελέσματα και επιδόσεις ε, σε τρέχοντα προγράμματα και είδαμε ότι παίρνουμε αποτέλεσμα σε 12 περιφερειές και 8 κράτη-μέλη συγκεκριμένα να χώρα αυτό το, αυτό το πείραμα και θα, τα αποτέλεσμα θα είναι έτοιμα σύντομα. Οι δείκτες που χρησιμοποιούμε στα τρέχοντα προγράμματα αποδεικνύεται ότι δεν περιγράφουν επαρκώς πολλές φορές τους στόχους των προγραμμάτων. Πολλές μάλιστα φορές βλέπουμε υπερβολικά μεγάλο αριθμό δικτών, σύγχυση για το περιεχόμενο του κάθε δίκτυ κλπ. Επίσης, διαπιστώνουμε ότι τα κράτη-μέλη πολύ συχνά δείχνουν έντονο ενδιαφέρον να μετακινηθούμε προ τα αποτελέσματα και τι επιδόσει. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα των δικτών, να υπογραμμίσω το εξή που είναι σημαντικό για την Κομισιόν. Θα πρέπει να απομακρυνθούμε από την οτροπία ότι οι δείκτε είναι κάτι τεχνικό και, και ότι μόνο ειδικοί και εμπειρογνώμονε είναι ικανοί να μιλούν για δείκτε. Όχι. Οι δείκτε θα πρέπει να περιγράφουν σωστά τι κάνει το κάθε πρόγραμμα. Και ένα μεγάλο κομμάτι συζήτηση για του δείκτε ε, είναι κοινή λογική. Εξετάζοντα του δείκτε των διαφορών προγραμμάτων, μελετώντας τους ε, λεπτομερώς ε, και το, και το τι πετυχαίνουν, ε, βλέπουμε, διαπιστώνουμε ότι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε πολύ το, πρόγραμμα, το, το σύστημα. Και ε, αυτός ο διάλογος θα πρέπει να γίνει και σε εθνικό και σε περιφερειακό και σε κοινοτικό επίπεδο. Θα πρέπει να δούμε πού θα δαπανούμε χρήματα, για ποιο λόγο, τι θέλουμε να αλλάξουμε, πώς μπορούμε να διαπιστώσουμε τι έχουμε πετύχει τους στόχους μας. Αυτές είναι οι ερωτήσεις που θα πρέπει να τροφοδοτήσουν τη συζήτηση. Τώρα, για το θέμα των κοινών δικτών και των ειδικών αναπρόγραμμα δικτών. Έχουμε κάποιους κοινού δείκτες και πρέπει να τους έχουμε έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε αθροίς και συγκρίσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να ενημερώνουμε και εσά τι γίνεται με την πολιτική μα. Σε ό,τι αφορά όμω του δείκτε αποτελεσμάτων, χρειαζόμαστε περισσότερου τέτοιου δείκτε ανά πρόγραμμα, έτσι ώστε να μπορούμε να μετρήσουμε τι αλλαγέ που επιδιώκει κάθε πρόγραμμα. Γιατί αυτέ οι αλλαγέ θα είναι διαφορετικέ ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο θα λειτουργούμε και θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις περιφέρειες και τα κράτη-μέλη να εντοπίσουν κάθε φορά λίγους κατάλληλους δείκτες επιδόσεων και να τους ε, παρακολουθούμε ε, ε, και να τους συζητούμε με την παράδοση του χρόνου. Τέλος να πω ότι στις συζήτηση που λαμβάνουν χώρα η Κομισιόν προετοιμάζει διάφορα δελτία που θα εξηγούν ορισμένα από τα στοιχεία για τα οποία μιλάμε σήμερα. Ε, αυτά τα δελτία θα φτάσουν και σε εσά. Φαντάζομαι ότι θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη στην τελική εκδοχή της έκθεσης. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το πλαίσιο επιδόσεων, γιατί υπάρχουν κάποιες παρανοήσεις για το τι, προτείνουμε, για το τι προτείναμε στις αρχικές μας προτάσεις. Το πλαίσιο επιδόσεων ε, έχει σχέση με την παρακολούθηση του κατά πόσον τα προγράμματα υλοποιούνται με βάση το σχεδιασμό τους, σύμφωνα με το σχεδιασμό τους και πιστεύουμε ότι εκεί θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία υπό τον έλεγχο των ε, αρχών διαχείρισης. Δεν θέλουμε, δεν επιδιώκουμε κανένας είδους ποινή ή κύρωση για στοιχεία και παράγοντες οι οποίοι δεν είναι υπό τον έλεγχο της αρχής διαχείρισης. Συνεπώς, ε, συγχαρητήρια για την μελέτη, θα τη διαβάσουμε λεπτομερώς, σύντομα και ελπίζω ότι θα ξανασυζητήσουμε αυτά τα θέματα σύντομα με την Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω άλλη μία αναφορά σε αυτά που μας ανέφερε μόλις η κυρία Πελεγκρίνο πριν κλείσω το θέμα αυτό. Το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι πριν από ένα χρόνο έγινε μια σχετική συζήτηση όπου κατέστησε σαφές ότι θέλουμε κάθε χρόνο όταν γίνεται η συζήτηση για την ε, απαλλαγή για τα σφάλματα των κρατών μελών, ότι παράλληλα θα πρέπει να γίνεται και μία συζήτηση στο Κοινοβούλιο για τα αποτελέσματα. Αν λοιπόν θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε τη συζήτηση των αποτελεσμάτων και των σφαλμάτων και να έχουμε τον σχετικό πίνακα, γιατί καταλαβαίνουμε ποια είναι η προστιθέμενη αξία για τον Ευρωπαίο πολίτη. Σας ευχαριστώ λοιπόν που τα τονίσατε αυτά τα θέματα περί του ρόλου του Κοινοβουλίου Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλό το ότι ακούσαμε τα απορίσματα. Μπορεί να μην συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 100% αλλά είναι εξαιρετικά χρήσιμο για μας στη φάση αυτή των ε, συζητήσεων και του επόμενου προγραμματικού επίπεδου. Και να περάσουμε στο επόμενο θέμα στην ατζέντα για το ρόλο της ε, πολιτικής συνοχής της ιδιαίτερα αποκρομισμένης περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Να ζητήσω από τους κοιόδες ιδιαίτερος να είναι πάρα πολύ σύντομοι γιατί δεν, δεν έχουμε όσο χρόνο θα θέλαμε και να δώσω το λόγο στον Νουνό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται. Η πολιτική συνοχής ε, παίζει σημαντικό ρόλο στις εξόχους απόγεντες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι προφανές. Θα πρέπει όμως να κάνουμε μια πολιτική επιλογή και να δεχτούμε ότι η πολιτική συνοχή είναι σημαντική για αυτέ τι περιοχέ για να επιτύχουν του στόχου στρατηγική Ευρώπη 2020. Γιατί το να θεωρήσουμε ότι είναι δυνατόν να επιτευχθούν αυτοί, αυτοί οι στόχοι χωρί επαρκή, επαρκή χρηματοδότηση είναι ουτοπικό. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια βιώσιμη, συμπεριληπτική και έξυπνη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό το λόγο δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε και την διάσταση των απόκεντρων περιοχών. Οι από απόκεντρες ε, περιοχές χαρακτηρίζονται από συνθήκες πολύ πιο δυσμενείς και γι' αυτόν τον λόγο η πολιτική συνοχή ιδιαίτερα σε αυτές τις ε, περιφέρειες θα πρέπει να έχει ε, να χρησιμοποιήσει εργαλεία, τα διορθωτικά ταμεία συγκεκριμένα, που να αυτά τα προβλήματα και αυτές τις συνθήκες να τις μετατρέψουν σε ευκαιρίες και να μειώσουν έτσι τις διαφορές. Η έκθεση την οποία σας υποβάλλω ε, χωρίζεται σε τρεις άξονες. Πρώτον, ε, ζητούμε μια διαφορετική ε, συμπεριφορά σε ό,τι αφορά αυτές τις περιοχές. Δεύτερος άξονας, όπου υποστηρίζουμε ότι χρειάζεται με ένα ιδιαίτερο πλαίσιο για τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ για τι εξόχου απόγεντε περιοχέ, με ιδιαίτερα μέτρα. Και τρίτον, μια καλύτερη διακυβέρνηση και συμμετοχή αυτών των περιφερειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί επειδή είναι ακριβώ απομακρυσμένε από το κέντρο, χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Αναλύοντα την πρόταση του πολιετούς ε, δημοσιονομικού πλαισίου, που θα το συζητήσουμε και στην επόμενη, στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης για το 2014-2020, ε, θα πρέπει να δώσουμε προσοχή σε συγκεκριμένα ζητήματα. Πρώτον, μεταξύ 2007-2013 ο προϋπολογισμός τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ήταν 975 δισεκατομμύρια ευρώ και για την περίοδο 2014-2020 προβλέπεται 1025 ε, δισεκατομμύρια. Ε, η πολιτική συνοχής περνάει από 347 σε 376 εκατομμύρια ευρώ συμπεριλαμβάνοντας και τα 50 ε, εκατομμύρια για, το, για, το, για την, ε, το ταμείο, τη δράση Connecting Europe. ο Με αυτόν τον τρόπο η πολιτική συνοχή ξεπερνάει την, ε, τον προπολογισμό τη γεωργική ε, πολιτική που από 416 περνάει στα 471 εκατομμύρια. Σε αυ... Οι περιοχέ συνοχή ε, είχαν 273 εκατομμύρια και θα περάσουν στα 162 εκατομμύρια ευρώ στην επόμενη περίοδο, 2014-2020. Αυτή η διαφορά, συγγνώμη, αυτές είναι οι περιοχές σύγκλησης ε, έχουν ξεπε... Ε, πολλές από αυτές τις περιοχές έχουν ξεπεράσει το 75% του μέσου ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπώς έχουν φύγει, γι' αυτό το λόγο έχουμε μείωση των ποσών. Αν εξετάσουμε τον προπολογισμό ε, των περιοχών ανταγωνιστικότητας και ε, ε απασχόλησης, περνάμε από τα 55 στα 53 εκατομμύρια ευρώ. Το είχα πει και σε προηγούμενη συνεδρίαση. Σας είχα υπογραμμίσει αυτή τη διαφορά. Έχουμε μια μείωση κατά 3%. Αν το συγκρίνουμε με, τις, με το προπολισμό για τις ε, ε, εξόχους απόκειτες περιοχές, έχουμε μία μείωση ε, η οποία ως ποσοστό είναι μικρότερη. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσω εγώ στους συμπολίτε μου πώς είναι δυνατόν οι πλούσιες περιοχές της Ευρώπης που έχουν ένα ΑΕΠ πολύ ψηλότερο από το μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βλέπουν τον προπολογισμό τους να μειώνεται 3% ενώ οι εξόχως κέντρες περιοχές, οι οποίες πολλές φορές είναι οι πιο φτωχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε μία μείωση 5 περίπου της Ε, όμως, ξεκινάμε από λαθασμένο σημείο. Γιατί συγκρίνουμε τα 976 με τα 926 και λέμε μείον 5%, αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Γιατί τα 976 συμπεριλαμβάνουν και τις αεροκατοικημένες περιοχές. Ενώ τα 926 της προηγούμενης περίοδου συμπεριλάμβαναν μόνο τις εξόχως απόγευτες περιοχές. Οπότε θα έπρεπε να συγκρίνουμε τα 976 με 1020 περίπου. Δηλαδή μιλάμε για μια διαφορά περίπου 40%. Οπότε θα πρέπει να του εξηγήσω πώ είναι δυνατόν οι εξόχου από τι περιοχέ να βλέπουν τον προπολογισμό να μειώνεται κατά 40% όχι κατά 5%. Και αυτό για σταθερέ τιμέ. Αν συγκρίναμε με τι τιμέ του 2011, θα έπρεπε να συγκρίνουμε τα νούμερα. 1.738 δισεκατομμύρια με 926 για την περίοδο 14-20. Μιλάμε λοιπόν για διαφορά 47% μείωση, περικοπή του προπολογισμού. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε λοιπόν. Γιατί δεν είναι κατανοητό πώς είναι δυνατόν η πρόταση της Κομισιόν να παραμελεί τόσο πολύ τις εξόχους τις περιοχές. Πώς είναι δυνατόν αυτές οι περιφέρειες να συμμετέχουν στη στρατηγική 2020, να την αναπτύξουν, να εφαρμόσουν την ε, έξυπνη ευφύ ανάπτυξη με τέτοιου είδους περικοπές. Η έκθεση αυτή ε, θα υποβληθεί Λίγο πριν η Κομισιόν υποβάλει τι ε, προτάσει τη ε, για τι ε, εξόχου απόκριτε περιοχέ, που θα, κάτι θα γίνει στο τέλο του πρώτου εξαμήνου. Γι' αυτό λόγο είναι ιδιαίτερα σημαντική η έκθεσή μα. Θα ήθελα να δούμε τι ακριβώ είναι το πιο σημαντικό. θα διατηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα έτσι ώστε η έκθεση να υιοθετηθεί στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια έγκαιρα έτσι ώστε να επηρεάσουμε το έργο της Κομισιόν, της εργασίας της Κομισιόν. Θα πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί ε, και να υποστηρίξουμε την αρχή της συνοχής, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις εξόχους απόγευτες περιοχές. Θα ήθελα τελειώνοντας να σας επιστήσω την προσοχή στο εξή. Ενημερώθηκα σήμερα ότι το έγγραφο που βρίσκεται στο ίντερνετ και που διανεμήθηκε στην αγγλική του εκδοχή έχει ορισμένα λαθάκια μεταφραστικά. Νομίζω ότι ήδη διορθώθηκαν και σας έχει διανεμηθεί μια καινούργια εκδοχή με τη σωστή μετάφραση. Αυτή να έχετε ως βάση παρακαλώ. Να ευχαριστήσω πολύ επίσης τη γραμματεία της ε, Επιτροπής που ακούραστα με βοήθησε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Είμαι στη διάθεσή σας να συζητήσουμε την έκθεση και βέβαια είμαι στη διάθεση των σκιωδών εισηγητών για να εργαστούμε μαζί σε τη βάση αυτού του κειμένου. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε υπεύθυνοι επιτροπή για θέματα που αφορούν τις υπερπεριφερειακές ε, και απόκεντρες περιοχές. Χαιρόμαστε για τη θέληση της Προέδρου, καθώς και του συναδέλφου του κ. Τεσέιρα, που επέτρεψαν τη σύνταξη αυτής της έκθεσης. Καταρχάς θα πρέπει να τονίσουμε την σημαντική δουλειά που έκανε ο εισηγητής μας για αυτό το θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ ευρύ. Είναι κρίμα που κάποιες μεταφράσεις, ε, όπως είπε και ο εισηγητής μας, ε, προδίδουν λίγο την προσπάθεια που έγινε και εμποδίζουν ορισμένους συναδέλφους ε, να συλλάβουν την ουσία του θέματος. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της έκθεσης, η πρώτη προτεραιότητά μας θα πρέπει να είναι η καταγγελία της μείωσης ε, των πιστώσεων για αυτές τις περιοχές. Είναι άδικο αυτές τις περιοχές να είναι οι μόνες οι οποίες αλλάζουν κατηγορία και μειώνονται οι που χορηγούνται σε αυτές. Εξ ονόματος της ομάδας έχω να υποβάλω ορισμένες τροπολογίες για να δούμε πού ακριβώς παρεμβαίνει η πολιτική συνοχής ε, στις περιοχές αυτές. Θα πρέπει να υπάρχει συντονισμό των παρεμβάσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όμω από την άλλη η ιδιαιτερότητα των ε, περιοχών αυτών, και νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει να έχουμε κριτήρια κατανομής των πόρων, ε, χρησιμοποίησης καινοτόμων μεθόδων χρηματοδότησης, ε, η σύναψη των ε, δημοσίων συμβάσεων και ιδίω. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει ανεπαρκής διασύνδεση αυτών των περιοχών. Την στιγμή που η Κομισιόν καταγγέλει την πρόσβαση των περιοχών αυτών στην ενιαία αγορά. Επίσης, θα πρέπει να συντονίσουμε καλύτερα τις εξωτερικές και εσωτερικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προτάσεις της Κομισιόν ενδιαφέρουσες, αλλά υπάρχουν προφανείς περιορισμοί. Γιατί η προσέγγιση είναι τεχνοκρατική και από πάνω προς τα κάτω. Εν είδη παραδείγματος, η Κομισιόν θέλει όλες οι χώρες εταίροι να επικυρώσουν την πρόταση για την εδαφική συνεργασία χωρίς να γνωρίζουν να έχει γίνει πλήρης εξέταση. Ο εισηγητής επίσης βασίστηκε στις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας και έκανε προτάσεις που δεν αφορούν μόνο την περιφερειακή πολιτική, αλλά αφορούν όλες τις δράσεις που μπορεί να προωθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ των περιοχών αυτών. Αλληλεία, έμπορο, ε, εμπόριο, ε, τελωνία κτλ. Αυτό που δημιουργείται για την Ευρωπαϊκή Ήπερο, λόγω του άρθρου 349 χρειάζεται μια ελάχιστη προσαρμογή, ούτως ώστε να είναι πραγματικά αποτελεσματικό στις απόκεντρες περιοχές. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε μια καινοτόμα προσέγγιση ε, και ερμηνεία αυτού του άρθρου, ούτω ώστε αυτέ οι περιοχέ να παίξουν πιλωτικό ρόλο στην Ευρώπη και να υπάρξει ένα καινοτόμο πειραματισμό σε ό,τι αφορά τι κοινοτικέ ρυθμίσει, να υπάρξουν πειραματισμοί οι οποίοι συνεχεία μπορούν να επεκταθούν και στην υπόλοιπη επικράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you. Is Η κυρία Γκρέσ είναι εδώ. Όχι. Ο κύριος, ο κύριος Χρυσόγελος. Yes. Ε, θα, ήθελα να... θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για την αψία της κυρία Κατρίν ε, δεν μπορούσε να έρθει και θα είμαι εγώ ε, ο μιλητής. Είναι η πρώτη φορά και θα με συγχωρήσετε για κάποιες ε, παρεμβάσεις. Ε, I have some remarks to say. In the local list of visas there is no reference να κάνω κάποια σχόλια. Δεν γίνεται αφορά σε μια σημαντική μελέτη για το ρόλο την, της πολιτικής συνοχής σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις εξόχως απομακρυσμένες περιοχές. Στο σημείο D θα ήθελα να αναφέρω να προτείνουμε μάλλον κάποια διατύπωση για την βιώσιμη γεωργία που θα πρέπει να αναφερθεί και να, να εφαρμοστεί στην εσωτερική αγορά. Στην παράγραφο 6 έχουμε επίσης μια ανάγκη προσθήκης για τις ε, συμφωνίες εμπορικής συμφωνίες με τρίτες χώρες. Οι χώρες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις στις απομακρυσμένες περιοχές. Στην παράγραφο 12 θα θέλαμε να υπάρχει μια αναφορά στην ενεργειακή αποδοτικότητα για την ε, παροχή κινήτρων σε ό,τι αφορά την κατανάλωση. Είμαστε υπέρ της καλύτερης διακυβέρνησης ε, στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να πάρουν χώρα, αν θέλετε, και το λόγο οι περιφέρειες για να ε, προτείνουν καλύτερους τρόπους διασύνδεσης. Εγώ προέρχομαι από μια τέτοια περιοχή με 38 νησιά από το Αιγαίο είμαι και σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των νησιών. Αυτά λοιπόν είναι απαραίτητα προκειμένου να συμμετάσχουν οι περιφέρειες αυτές στην ε, διαδικασία της Ευρωπαϊκής αναποίησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και η Πρόεδρος. Για... Θα συμφωνήσουμε σε λίγο για την προθεσμία για τις τροπολογίες που θέλετε να καταθέσετε. Ο κύριο Βλάσεκ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, να καλωσορίσω καταρχάς ε, κάποιες από τις προτάσεις της έκθεσης σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την ε, ενθάρρυνση και την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας των ε, απομακρυσμένων περιοχών σε ό,τι αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη μέσω των δικτύων υποστήριξη της καινοτομίας προκειμένου να περιοριστεί η εξάρτηση από την παραδοσιακή γεωργία. Ωστόσο, έχω και πολλές ανησυχίες να εκφράσω σε μια εποχή οικονομικής λιτότητας υπάρχει ανάγκη αποταμίευσης και περικοπής των προϋπολογισμών και στο πολιτές ε, χρηματοοικονομικό πλαίσιο τα ποσά που χορηγούνται στις εξόχως απομακρυσμένες περιοχές περιορίζονται για την περίοδο 14 έως 20. Και αυτό αποτελεί και τη δική μας θέση. Επίσης, δεν μπορούμε να αποτεχτούμε την ενίσχυση των μέτρων χρηματοοικονομικής υποστήριξης για τέτοια ζητήματα, όπως προτείνει η έκθεση. Το ECR πιστεύει ότι το οικονομικό μέλλον, μέλλον των περιοχών αυτών εξαρτάται από το εμπόριο, όχι από τις ε, αύξηση των επιδοτήσεων και δεν ε, επιλέγουμε την παράταση της ΚΑΠ. Και επίσης φαίνεται ότι επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά στις ε, νησιωτικές περιοχές. Γιατί να έχουν ιδιαίτερα ωφέλη αυτές οι νησιωτικές ε, περιοχές παρά το γεγονός ότι όλες ε, οι χώρες μέλη έχουν απομακρυσμένες περιοχές που χρήζουν συγκεκριμένης προσοχής. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τον Νούνο Τεσέιρα για την ποιότητα της δουλειάς του. Θέλω να του πω ότι συμφωνώ επί της ουσίας με τους βασικούς προσανατολισμούς και με τις βασικές προτάσεις που κάνει στην εκθεσή του. Είναι μια έκθεση που φτάνει την κατάλληλη χρονική στιγμή για δύο λόγους. Καταρχάς, λίγο, λίγους μήνες ή λίγες εβδομάδες πριν από τη νέα ανακοίνωση της, Επιτροπής για τις α, εξόχως απόκεντρες περιοχές. Και οι προτάσεις στην έκθεσή του νομίζω ότι θα είναι ένα σημείο, ένα στοιχείο που θα εμπνεύσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανακοίνωσή της. Φτάνει λοιπόν πολύ επίκαιρα για αυτόν τον πρώτο λόγο, αλλά και για ένα δεύτερο λόγο. Για την κρίση που πλήττει αυτή τη στιγμή το σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο τη κρίση, τη γενικευμένη κρίση, είναι σημαντικό η Επιτροπή μα, αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επαναδιατυπώσουν την υποστήριξή τους προς τις περιοχές αυτές που λόγω του ευάλωτου της οικονομίας τους, λόγω της εξάρτησής του, από το εξωτερικό, λόγω της απομάκρυνσής τους από τις αγορές είναι οι πρώτες που πλήττονται από την κρίση. Από αυτή την άποψη δίκιο έχει ο εισηγητής που τόνισε την ανάγκη να διατηρήσουμε ένα κατελάχιστο στα ίδια επίπεδα της πιστώσης και για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού ε, και μάλιστα να υπάρξει μια αύξηση των, ε, της πρικοδότησης, της χρηματοδότησης των ΠΟΖΕΗ. Όλοι οι ομιλητές που μίλησαν είπαν ότι υπάρχει πρόβλημα με τις πιστώσεις αυτές που θέλουν να αντισταθμίσουν την αύξηση του κόστους, ή μάλλον το αυξημένο κόστος. Εμεί ε, ε, ήμουνα μέλος της αντιπροσωπείας που έθεσε ερωτήσει προς τον Επίτροπο Χαν. Ε, το ρωτήσαμε για ποιους λόγους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μία μείωση της χρηματοδότησης πάνω από το 40% είναι η μείωση αυτή. Για ποιο λόγο και ο Επίτροπος δεν μου απάντησε. Νομίζω ότι είναι σημαντικό όλοι οι ευρωβουλευτές της Επιτροπή μας θα πρέπει να πιέσουν, την, να πιέσουν ακόμα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ακρίβεια της ζωής και το επιπλέον κόστος είναι ε, ένα χαρακτηριστικό που το βλέπουμε σε όλες αυτές τις περιοχές. Η έκθεση που παρήγγειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πιστοποιεί ότι υπάρχει παντού αυξημένο κόστος. Ε, ήρθα σήμερα το πρωί από, την, ε, από το νησί Ρεϊνιόν ε, ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει κρίση εκεί, λόγω της ακρίβειας της ζωής, λόγω της εξάρτησης από το εξωτερικό και λόγω των προβλημάτων της τιμής της ενέργειας και των πρώτων υλών και των, και των ειδών διατροφής. Όλα αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το επιπλέον κόστος, η αύξηση του κόστους. Και τελειώνω με το θέμα της ενέργειας, που είναι το κλειδί της ανάπτυξης των περιοχών αυτών. Θέλω να μιλήσω ειδικά για τις ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας. Ξέρω ότι αναφέρονται στην έκθεση του συναδέλφου και τα νησιά αυτά λόγω της γεωγραφικής τους θέσης μπορούν να πετύχουν ένα πιο φιλόδοξο στόχο από άλλες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο στόχος της ενεργειακής αυτονομίας δεν είναι ένας ε, δεν είναι ένα στόχο ο οποίο δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Αντίθετα. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επαναλαμβάνω και εγώ τα συγχαρητήρια ε, στο, προς τον κύριο Τεσέιρα. Η έκθεση αυτή πραγματικά περιλαμβάνει όλες τις ε, προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτές οι περιοχές. Επίσης περιλαμβάνει η έκθεση πολλά από τα επιχειρήματα του κοινού Memorandum Γαλλίας-Ισπανίας-Πορτογαλίας ε, ε, που υποβλήθηκε επί Ισπανικής Προδίας του 2010 καθώς επίσης στην έκθεση Σόλμπες και, στην, και, από, τα, ε, και από την συνάντηση των αξόχων περιφερειακών περιοχών που έλαβε χώρα στη Μαρτίνικα του 2011. Είναι σίγουρο ότι χρειάζεται ιδιαίτερη μεταχείριση αυτών των περιοχών, των περιφερειών. Επίσης είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε διαφορετικά κριτήρια και όχι το κατακεφαλήν ΑΕΠ. Αυτό το κριτήριο δεν επαρκεί για να περιγραφεί η κατάσταση των περιφερειών αυτών. Χρειάζονται και άλλοι δείκτες όπως η ανεργία, η ανεργία των νέων ε, και το ποσοστό προώρης εγκατάλειψης της σχολικής εκπαίδευσης. Επίσης είναι σημαντικό να αυξηθεί η κοινοτική συγχρηματοδότηση ιδιαίτερα για τα εργαλεία στήριξης. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε αντιθέτως μια μείωση του συνολικού προπολογισμού κατά 40%. Ε, επίσης η αντιστάθμιση ε, το, του υπερκόστους στο ποσέι αλίας για τη δημιουργία μιας πραγματικής οικονομίας ε, της θάλασσας και της αλίας. Χρειάζεται επίσης να συμπεριλάβουμε μια αναφορά στην ανάγκη να αξιολογηθεί, να αξιολογείται κάθε φορά ε, από τεχνικής πλευράς ο αντίκτυπος οποιασδήποτε συμφωνίας που γράφεται με τρίτες χώρες πριν αυτή η υπογραφή. Έτσι ώστε να προσδιορίζεται ο αντίκτυπος και να εντοπίζονται τα κατα... οι κατάλληλες αποζημιώσεις και αντισταθμίσεις. Ε, επίσης, ε, η, ε, είναι απαραίτητο να έχουμε ένα συγκεκριμένο κριτήριο χρηματοδότηση ανεξαρτήτως της απόστασης. Δεν συμφωνώ όμως με την πρόταση του κ. Τεσέρα να χρησιμοποιηθούν άλλα κριτήρια ε, για την κατανομή των πρόσθετων πιστώσεων του ΦΕΝΤΕΡ. Ο συνολικός πληθυσμός της κάθε περιφέρειας νομίζω ότι είναι το πιο κατάλληλο κριτήριο. Θα υποβάλω και κάποιες συγκεκριμένες τροπολογίες. Ευχαριστώ. Λουίς Ευχαριστώ. Δύο λόγια μόνο. Η έκθεση αυτή είναι πολύ επίκαιρη και κέρια γιατί μέσω των διασκέψεων των ε, Πρόεδρων ε, έχουμε επαρκή στοιχεία η Κομισιόν γνωρίζει το θέμα είναι έτοιμη να υποβάλει τις προτάσεις της, έχει την έκθεση Σόλμπε στα χέρια της. Αυτή η πρωτοβουλία θα επιτρέψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν την υποβολή των προτάσεων της Κομισιόν να κάνει γνωστή τη δική του θέση. Ο Νούνο Τεσέιρα παρουσίασε πολύ σωστά τα βασικά προβλήματα τη δυσκολία συμμετοχή στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκή τη δυσκολία αυτών των περιφερειών ε, στην ε, περιφερειακή ενοποίηση. Είμαστε απομακρυσμένες περιοχές από την Ήπειρο, από το κέντρο. Ο Νούνο πολύ σωστά τα περιγράψε όλα αυτά. Η νέα αρχιτεκτονική της πολιτικής συνοχής ε, θα είναι νομίζω μια ενδιαφέρουσα μέθοδος για την, τον καθορισμό μια κοινωνικής στρατηγική και για τις εξόχω περιφερειακές περιοχές, περιφέρειες. Χρειαζόμαστε επιχειρησιακά προγράμματα για συγκεκριμένους ε, τομεί και μια γενικότερη πολιτική για όλες τις περιοχές και για όλους του τομείς. Θα πρέπει ε, ε, η πολιτική αυτή να βοηθήσει αυτές τις περιφέρειες να εκμεταλλευτούν όλο τους το δυναμικό. Θα ε, υποβάλλουμε και κάποιες τροπολογίες. Ευχαριστώ. Good Thank you very much. Ευχαριστώ. Το βασικό μήνυμα της έκθεσης αυτής του εισηγητή μας είναι γιατί υπάρχουν τόσο έντονες περικοπές. Γιατί με βάση τα νούμερα που είπε η περικοπή αυτή είναι 40%. Εγώ δεν, δεν το είχα καταλάβει αυτό. Τα νούμερα δεν είναι ξεκάθαρα. Μέχρι να μας δώσει η Κομισιόν μια πραγματική απάντηση θα υπάρχουν προβλήματα. Στην πρώτη συνεδρίαση που κάναμε φέτος, το 2012, είχαμε τον Επίτροπο δίπλα σας. Εγώ το έδωσα ένα πίνακα. Και όπου ε, βλέπαμε ότι ότι για την πολιτική συνοχή στην πραγματικότητα η περικοπή είναι μείον 20% η περικοπή των πιστώσεων. Επίσης, τι πιστώσεις θα έχουν η κάθε κατηγορία περιοχών, οι ανεπτυγμένες, οι λιγότερο ανεπτυγμένες και οι εξόχως απόκεντρες. Πριν από τέσσερι εβδομάδε τον ρώτησα τι περικοπέ θα υπάρχουν για κάθε κατηγορία, αλλά δεν μου απάντησε. Αν δεν έχουμε χρήματα στην Ευρώπη, φυσιολογικό είναι να, να περικόψουμε. Αλλά τότε θα πρέπει να εξηγήσουμε σε όλα τα μέλη τη Επιτροπή, να μα εξηγήσει η Επιτροπή δηλαδή, πώ γίνονται αυτέ οι περικοπέ. Και καλύτερα θα τα μα τα εξηγήσει όλα αυτά γραπτό. Να μα εξηγήσει τα νούμερα. Πριν από ένα μήνα, το μόνο που μου είπε η Επιτροπή ήταν κάτι γενικό χωρίς νούμερα. Αυτό είναι πρόβλημα, έτσι. Και δεν αφορά μόνο τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίσαμε και εμείς εδώ, αλλά θα υπάρξουν και τέτοια προβλήματα και σε άλλες εκθέσεις, σε άλλες ε, ε, επιτροπές. Δεν καταλαβαίνω πώς μερικές φορές στις πιστώσεις πληρωμών έχουμε αυξήσεις, αλλά εδώ πέρα προβλέπονται τέτοιες μεγάλες περικοπές. Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για την λογική. Θα πρέπει να μας εξηγείτε και τα νούμερα. Να μας λέτε τόσα για, αυτή τις, για αυτές τις περιοχές, τόσα για τις άλλες. Το βασικό ερώτημα που θέτει ο εισηγητή δεν μπορούμε να το απαντήσουμε. Λέει ότι οι πιο απομακρυσμένε περιοχέ θα υποστούν μείωση σε 40%. Εγώ δεν το πιστεύω γιατί μου φαίνεται τεράστια αυτή η περικοπή. Μα το λέει, αλλά εμεί δεν έχουμε τίποτα να το αντιτάξουμε γιατί δεν μα έχει δώσει κανένα στοιχείο η Γενική Διεύθυνση, η Ρέτζιο ή οποιοδήποτε άλλο. Όσο δεν μα δίνει νούμερα θα έχουμε πρόβλημα. Ε, Έχουμε ως επόμενο σημείο το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Ε, Χρειαζόμαστε τα νούμερα. Δεν μπορούμε να λέμε «Α, δώστε μας χρήματα». Πρέπει να ξέρουμε αν για τις ε, περιοχές μετάβασης να έχουμε 47% αύξηση, για τις ανεπτυγμένες περιοχές συν 4% αύξηση των πιστώσεων, και για τις εξόχους απόκεντρες μείω 40. Είναι δυνατόν. Όσο δεν ξέρουμε τα νούμερα, όλα τα υπόλοιπα είναι φλιναθήματα. Ευχαριστώ. Ο Νούνο. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω λίγο τα πράγματα και να ξεκινήσω με το εξής. Ε, είναι πολύ σωστό ότι ε, τα νούμερα τα οποία υποβλήθηκαν ακόμα και στην Επιτροπή Προεπλογισμού δεν είναι σωστά. Διότι ε, οι πληροφορίε που έλαβε συνάδελφο δεν ήταν σωστέ. Και εγώ υπέβαλα γραπτό ερώτημα στην Κομισιόν για αυτά τα νούμερα του ΦΕΝΤΕΡ, του προεπλογισμού του ΦΕΝΤΕΡ. Και η Κομισιόν μου είπε ότι υπάρχουν λάθη στα στοιχεία τα οποία μου είχαν δοθεί. Τώρα έλαβα τις πληροφορίες ότι τα, αυτά τα συγκεκριμένα νούμερα που σας παρουσίασα είναι τα σωστά. Δηλαδή, επιβεβαιώνω ότι οι μειώσεις του ΦΕΝΤΕΡ για τις αξιόχως περιφερειακές περιοχές και τις αεροκατοικημένες περιοχές ε, των βορείων ε, ε, περιοχών ε, είναι 47%. Ε, από 1738 εκατομμύρια περνάμε στα 926 εκατομμύρια μεταξύ της προηγούμενης και της ε, επόμενης ε, περίοδου 2014-2020. Συμφωνώ με επίσης με τον κύριο Βλόσακ. Δεν θέλω να μείνετε με την λαθασμένη ιδέα ότι οι εξόχως κομμακρισμένες περιοχές είναι ε, ένα πράγμα. Ε, η Γαλλική Γουιάννα είναι η μόνη περιοχή η οποία δεν είναι από αυτές. Ε, αλλά βρίσκεται στα 10.000 περίπου χιλιόμετρα από την Ευρώπη, έτσι κι αλλιώς. Καμία από αυτές τις περιοχές δεν θέλει να επιβιώσει για το υπόλοιπο της ιστορίας ε, ει βάρος του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Όχι. Ε, η αρχή της ισότητας όμως ε, μας λέει ότι θα πρέπει να συμπεριφερθούμε με τον ίδιο τρόπο σε αυτούς που είναι ίσοι μεταξύ του και με διαφορετικό τρόπο σε αυτούς που είναι διαφορετικοί. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να συμπεριφερθούμε με τον ίδιο τρόπο σε μια περιοχή, η περιφέρεια που βρίσκεται στο κέντρο τη Ευρώπη, στον πυρήνα τη Ευρώπη. με ε, μια περιοχή η οποία βρίσκεται 10.000 χιλιόμετρα μακριά ε, είναι ένα νησί όπως η Γουαδελούπη ή η Γαλλική Γουιάννα. Συνεπώ δεν είναι δυνατόν να συγκρίνουμε πράγματα τα οποία δεν είναι ομοειδή. Η Γαλλική Γουιάννα ασφαλώς θα ήθελε να επιβιώσει χάρη στο εμπόριο. Να σας δώσω ένα σαφές παράδειγμα πως η πολιτικές λιτότητας έχουν χρησιμοποιηθεί, έχουν εφαρμοστεί σε αυτές τις περιοχές. Στη Μαδέιρα, από όπου προέρχομαι εγώ, όπως γνωρίζετε, η Πορτογαλία βρίσκεται μέσα σε ένα πρόγραμμα διάσωση, πολιτική λιτότητας, χρηματοδοτούμαστε από την ε, Τρόικα, ε, Κομισιόν Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, Δουνουτού κλπ. Μπορούμε να πούμε το εξή ότι στον επόμενο προπολογισμό της Μαδέιρα Ε, έχουμε, ο επόμενος προπολογισμός θα είναι 126 εκατομμύρια ευρώ. Το 2011, εξαιτίας της διακοπής του φορολογικού καθεπροτιμησιακού καθεστώτος της ε, Μαδέιρα, εξαιτία των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα, έχασε η Μαδέιρα 140 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς μπορούν να επιβιώσουν αυτόνομα, αλλά θα πρέπει να βοηθηθούν αυτές οι περιοχές. Επίσης μην ξεχνάμε ότι ο συγκεκριμένος προπολογισμός δεν αφορά μόνο τις αξόχως ε, απομακρυσμένες περιοχές. Πολύ συχνά εστιαζόμαστε σε αυτές. Αλλά μερικές φορές ξεχνάμε τις αεροκατοικημένες περιοχές των ε, χωρών της ε, ε και των βόρειων χωρών, πιο συγκεκριμένα. και υπάρχει κάποια, ε, κάποια αντίφαση. Δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν η πρόταση Κομισιόν για το ΦΕΝΤΕΡ στο 11ο άρθρο να αναφέρει ε, ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη προϋπόθεση, μια αρεσιμότητα ε, και λέει το 50% των πόρων θα πρέπει να αφιερώνεται στις θεματικές ε, συγκεντρώσεις για τις ε, εξόχους περιφερειακές απομακρυσμένες περιοχές, αλλά δεν αναφέρει τίποτα για τις αεροκατοικημένες περιοχές των βορείων χωρών. Συνεπώς, σίγουρα δεχόμαστε ότι θα πρέπει να γίνουν θυσίες, περικοπές, αλλά ζητώ αυτές οι θυσίες να είναι δίκαιες. Δεν είναι δυνατόν να μειώνουμε 3% τον προπολογισμό των πιο πλούσιων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 47% τον προπολογισμό των πιο φτωχών περιοχών. Είναι πολύ εύκολο, λέμε, στην Πορτογαλία να είμαστε ισχυροί με τους αδύνατους ε, από ότι αδύνατοι με τους ισχυρού. Θα πρέπει να κλείσουμε τη συζήτηση, αλλά νομίζω ότι ο Λάμπερτ Φανίστελ Ρόι θα να πάρει το λόγο εν συντομία. Ναι, ένα μικρό σχόλιο από πλευρά μου προς τον εισηγητή για όλους όσους θέλουν να καταθέσουν και τροπολογίες. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πρόκειται για ίδια πρωτοβουλία για τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την φιλοσοφία της πολιτικής για το 2020 σε ό,τι αφορά τις άκρως απομακρυσμένες περιοχές δεν ε, πρόκειται για ένα έγγραφο στο οποίο μπορούμε να ξεκινήσουμε μία μεγάλη συζήτηση για τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές. Άκουσα τις παρατηρήσεις σας, αλλά, αλλά ας εξετάσουμε και ποιες είναι οι στόχοι, ποιοι είναι οι στόχοι α, της έκθεσης ίδιας πρωτοβουλίας για να μην καταθέσουμε ένα σωρό τροπολογίες για χρηματοοικονομικά ζητήματα τα οποία δεν μπορούν να μπουν σε αυτό το έγγραφο. Αυτός παρατηρήσει, επιτρέψτε μου. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος και η αναπαλλαλέηση που είναι διευθύντρια τμήματο, δεν θα της δώσουμε το λόγο, αλλά θα τη ζητήσουμε να μεταβιβάσει το μήνυμα αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ότι χρειαζόμαστε με την Επιτροπή μια συνάντηση για να διευκρινίσουμε αυτές τις δυσκολίες. Για να αποφασίσουμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν τώρα και αυτό που είπε ο Λάμπερτ είναι πάρα πολύ σαφές, δεν χρειάζεται να το επαναλάβω, σας ευχαριστώ. Αυτό που θα πρέπει να κάνω είναι να θέσω την ε, προθεσμία για τις τροπολογίες. Προτείνω 1η Μαρτίου στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Σας παρακαλώ συνάδελφοι λοιπόν να σεβαστείτε αυτή την προθεσμία. Και τα θέματα χρηματοδότησης θα τα συζητήσουμε και σε μελλοντικέ συζητήσεις. Και το θέμα των εξόχω ε, απομακρυσμένων περιοχών θα το ξαναδούμε. Μπορούμε να περάσουμε λοιπόν στην έκθεση την γνωμοδότηση Κοβάτσεφ ε, για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020. Έχουμε επί της ουσίας την Επιτροπή Προϋπολογισμού και τις εισηγητές ε, Μπέγκελ και καλφέν, Δεν θα γίνει σήμερα η συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Έχουμε τέτοιες ευκαιρίες στο μέλλον. Ε, θέλουμε να ακούσουμε απλά τους συζητητές για το πώς θα διαμορφωθεί η διαδικασία τους επόμενους μήνες. Δεν ξέρω, θέλει ο Άντρα να ξεκινήσει την παρουσίαση εν συντομία και μετά να ακούσουμε και τους εισηγητές. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε σήμερα να ανταλλάξουμε ιδέες σε ό,τι αφορά τον κανονισμό αυτό για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Την προηγούμενη φορά συζητήσαμε την διαδικασία συνένεση στο άρθρο 312 της συνθήκης που δεν επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να πει παρά μόνο ένα ναι ή ένα όχι στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό τι σημαίνει ότι εξαρτώμαστε πάρα πολύ από τα βήματα που λαμβάνει η Επιτροπή ε, Προϋπολογισμού, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ενδιάμεση έκθεση που καταθέτει βάση του άρθρου 81 του κανονισμού. Χαίρομαι που είναι εδώ οι δύο συνεισηγητές, αλλά εξ όσων γνωρίζω η Επιτροπή Προπολογισμού δεν έχει λάβει μια οριστική απόφαση και αυτό ε, δυσκολεύει το έργο των ε, συμβουλευτικών επιτροπών. Να αναφέρω ότι συναντήθηκα με τον κύριο Έρικ Φομπρέσκε από την Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συζητήσαμε πώς έχει η κατάσταση στο Συμβούλιο. Εστιαστήκαμε ιδιαίτερα σε θέματα εντολής διαπραγμάτευσης στις σχετικές επιτροπές. Έχουμε τους φίλους της Προεδρίας, την ομάδα αυτή εργασίας που εξετάζει πτυχές ε, της νομοθετικής πολιτικής, για παράδειγμα το πακέτο συνοχής, το πακέτο κοινή αγροτικής πολιτικής και όλες τις οικονομικές επιπτώσεις. Ενώ η άλλη ομάδα εργασίας θα εξετάσει άλλα ζητήματα όπως η θεματική συγκέντρωση για παράδειγμα. Ωστόσο, στη συζήτηση με τον, με τον κύριο Φομπρέσκα κατέστη σαφές ότι δεν υπάρχει μία σαφής γραμμή μεταξύ των δύο ομάδων εργασίας. Ε, ένα πλαίσιο διαπραγμάτευσης το οποίο προτίθεται να παρουσιάσει η Προεδρία Ιδανική τον Ιούνιο θα αποτελέσει τη βάση των συζητήσεων και ελπίζουμε τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν για το πλαίσιο αυτού των διαπραγματεύσεων. Κάτι που θα ήθελα να αναφέρω σχετικά με τα ποσά. Η Επιτροπή μας θεωρώ θα πρέπει να ενθαρρυνθεί να εξετάσει τα ποσά που α, εκχωρούνται σε κάθε πολιτική σύμφωνα και με την εκθέση Γκαρίγκα. Ξέρω ότι γίνεται μια τέτοια συζήτηση να μην παρουσιαστούν τα σχετικά ποσά, αλλά νομίζω ότι προκειμένου να ακουστεί η φωνή μας θα πρέπει να ζητήσουμε τέτοια συζήτηση. Και πάλι χαίρομαι που βρίσκονται εδώ και οι δύο συνεισηγητές και προσβλέπω να τους ακούσω. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι, ναι, αποφασίστε εσείς που θα ξεκινήσει. Αλφαβητικά, ο Ράιμερ Μπέγκε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι είμαστε καλοί σύμμαχοι ακόμα και αν προερχόμαστε από διαφορετικές ομάδες, γιατί νομίζω ότι είναι σαφές. Αν το Κοινοβούλιο στη διαδικασία έγκρισης για το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο θέλει να περάσει γνώμη του για τέτοια θέματα, αυτό θα το πετύχουμε μόνο από κοινού. Το ίδιο ισχύει και για το θέμα των νομοθετικών διαδικασιών και του διαδικασία του προπολογισμού. Μόνο από κοινού μπορούμε κάτι να πετύχουμε. Σε μια χρονική στιγμή, μάλιστα, που το συνολικό πολιτικό πλαίσιο δεν είναι τόσο απλό. Προκειμένου λοιπόν να περάσει αυτά που ψήφισε το, η Ολομέλεια βάσει της έκθεσης ΣΟΥΑ με την έκθεση, με συγκητή τον Σαλβατόρ Καρίγκα. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό πλαίσιο η Επιτροπή Προϋπολογισμού είναι αρμόδια για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και σε ό,τι αφορά τα έσοδα και σε ό,τι αφορά τις δαπάνες και σε ό,τι αφορά την πολιτική συνοχή είναι αρμόδια και η Επιτροπή σας. Θα κοιτάξουμε και θα πρέπει να συζητήσουμε πώς θα πρέπει να γίνει ο συντονισμός με σωστό τρόπο εδώ πέρα στο Κοινοβούλιο. Ξεκινήσαμε με τις δεσμεύσεις της Ουγγρικής Προεδρίας, μετά με το πρώτο εγχείρημα, αν θέλετε, με την ε, με το πρώτο απόπειρα με την Πολωνική Προεδρία και τώρα με την Δανική Προεδρία προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε την οδό μιας πιο συντατική ε, συζήτησης, ενό πιο συντατικού διαλόγου. Και αυτό προαπέτησε ε, δέσμευση και κάποια, ε, αν θέλετε, πίθο προς το Συμβούλιο και Όντω, βάσει του άρθρου 312 της συνθήκη της Λισαβόνας, σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό πλαίσιο των πολιτέ, έχουμε μια διαδικασία έγκριση. Άρα στο τέλο, μόνο ναι ή όχι μπορούμε να πούμε. Και αυτό το τονίζω. Μόνο ναι ή όχι μπορούμε να πούμε ως Κοινοβούλιο, αλλά παράλληλα στο άρθρο 312 παραγράφος 5 περιέχεται και μια διατύπωση που αναφέρει ότι το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διευκολύνουν την έγκριση των προτάσεων αυτών. Και αυτό οδήγησε σε μία μακρά νύχτα, αν θέλετε, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, που προσπάθησαν ε, οι υπεύθυνοι να παραγωνίσουν το Κοινοβούλιο. Καταφέραμε αυτό να το αποτρέψουμε σε ένα βαθμό. Θα πρέπει όμως ε, το πνεύμα αυτής της ε, συμφωνίας να εκπληρωθεί. Θα πρέπει προς το Συμβούλιο να απευθύνουμε μια προειδοποίηση. Να χρησιμοποιηθούν όλες οι δυνατότητες που έχουμε προκειμένου μέχρι τον Μάρτιο, μέχρι τον Ιούνιο να μπούμε σε πραγματικές διαπραγματεύσεις και όχι σε μια ευγενική ανταλλαγή απόψεων. Γιατί τότε όντως θα είναι δύσκολο να συγκεντρωθεί πλειοψηφία εδώ στο Κοινοβούλιο για την υποστήριξη του πολιτού του Ισλαμικού πλαισίου. Δεν θα ασχοληθεί μόνο με αριθμητικά στοιχεία αυτό το θέμα, αλλά και με τα μικρά γράμματα σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό. Αυτά λοιπόν που σήμερα που συμπεριλαμβάνονται σήμερα στην θεσμική συμφωνία, στην διεθνική συμφωνία, τα οποία όμως έχουν και μεγάλη πολιτική βαρύτητα. Καταρχάς, το ερώτημα της διαμόρφωσης του προϋπολογισμού, θέματα ευελιξίας εντός του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου και ούτω καθεξής. Και εμείς επιμένουμε να πετύχουμε σε ό,τι αφορά την προετοιμασία του διαπραγματευτικού πλαισίου που σκοπεύει να προετοιμάσει η Δανική Προεδρία, να εισέλθουμε σε μια φάση έντονου διαλόγου, προκειμένου τέτοιες βασικές προτάσεις να, σε τέτοιε βασικέ αποφάσει να ληφθεί υπόψη απαρκώ η άποψη του Κοινοβουλίου. Αυτά που μπορούμε να σα παρουσιάσουμε εμεί οι δύο σε αυτή τη φάση δεν είναι αποφασισμένα ω γραμμή, γιατί θα υπάρξει μια ομάδα εργασίας, ε, μια ομάδα επαφής από τους συντονιστές όλων των επιτροπών με τον πρόεδρο Σούλτς και εξ όσων διάβασα θα συμμετάσχουν κάποιοι πρόεδροι κάποιων σημαντικών επιτροπών την Τετάρτη προκειμένου να παρουσιάσουν τις απόψεις τους. Ε, οι δύο εισηγητές λοιπόν ε, έχουμε δηλώσει ότι θέλουμε να διεξάγουμε έναν δομημένο διάλογο τους επόμενους μήνες προκειμένου όλοι να γνωρίζουν τι γίνεται και επίσης την Ολομέλεια του Στρασβούργου την ε, Πέμπτη το απόγευμα να διοργανώνεται μία συζήτηση μεταξύ των συνεισηγητών προκειμένου να υπάρχει μια διαρκής ε, ανταλλαγή απόψεων προκειμένου να είμαστε όλοι ενήμεροι ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον. Και αυτό θα συζητηθεί σε λεπτομέρεια την Τετάρτη, αλλά εμείς όσοι συνεισηγητές ε, το έχουμε συμφωνήσει και θέλουμε να το προτείνουμε, θα πρέπει να προετοιμαστούμε για την Ολομέλεια του Μαΐου, ανάλογα με την πρόοδο των πραγμάτων, για να παρουσιάσουμε ένα ψήφισμα στην Ολομέλεια, που θα περιλαμβάνει διευκρινήσεις, αν θέλετε, και κόκκινες γραμμές από πλευράς του Κοινοβουλίου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στα πλαίσια των όσων έχουν ήδη υπερψηφιστεί στην ε, έκθεση Γκαρίγκα. Δεν χρειάζεται να τα ξανασυζητήσουμε αυτά, όταν τα επανεφαρευρούμε. Επιπλέον, θα πρέπει να σκεφτούμε στην πάροδο του χρόνου στις αρχές Οκτωβρίου κατά πάσα πιθανότητα, μήπως θα πρέπει να παρουσιάσουμε μια διάμεση έκθεση προτού προκύψει μία κατάσταση στο Συμβούλιο σε ό,τι αφορά τα αριθμητικά στοιχεία και τα άλλα πακέτα, γιατί ξέρουμε πώς πάνε τα πράγματα εκεί στο Συμβούλιο. Ίσως θα μπορούσαμε λοιπόν να ζητήσουμε εντολή από την όλη μέλεια, προκειμένου να εκφράσουμε την απόψή μας σε μία ενδιάμεση αξιολόγηση, σε μία ενδιάμεση έκθεση, σε θέμα των αριθμητικών στοιχείων, σε ό,τι αφορά τα νούμερα. Ξέρω ότι γίνεται στις διάφορες ομάδες μια ξεχωριστή συζήτηση. Να σας επενθυμίσω το εξή, ωστόσο. Το 2005 έγινε μια συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων προκειμένου όλα τα θεσμικά όργανα να δεσμευτούν να επιτελούν το έργο τους συμπεριλαμβανομένης του καθήκοντος για παράδειγμα της πρώτης ανάγνωσης αλλά να μην ορίζονται οριστικά αριθμητικά στοιχεία αλλά στο τέλος μόνο βάσει της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συζητιέται το πώς θα κατανέμονται τα ποσά αυτά. Ξέρω ότι υπάρχουν και άλλες απόψεις. Ε. Ξέρω ότι κάποιοι έχουν πρόβλημα να παρουσιάζουν ποσά. Να θυμάστε όμως το τι θα προκαλέσει αυτό εδώ στο Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την πολιτική συνοχή και την πολιτική αγροτική ανάπτυξης έχουμε σαφείς ε, ε, διατυπώσει. Στο κεφάλαιο 67, για παράδειγμα, της πολιτικής συνοχής αναφέρεται ότι τα ποσά ε, τα οποία είχαν προταθεί και είχαν αποφασιστεί στην προηγούμενη πραγματική περίοδο θα πρέπει τουλάχιστον να διατηρούνται στην επόμενη περίοδο και το καθεξής. Αυτό τι σημαίνει ότι υπάρχει ένα περιθώριο ελιγμού και για άλλους ε, πολιτικούς ε, τομείς όπου υπάρχει ένας αυτόματος δείκτης ε, πληθωρισμού 2% αυτό αποτέλεσε συμβιβασμό. Αν τώρα ξεκινήσουμε σε κάθε, σε κάθε νομοθετική πρόταση να αναφέρουμε ποσά, Ίσως στο θέμα της πολιτικής συνοχής και στο θέμα της αγροτικής ανάπτυξης να είναι πιο εύκολα τα πράγματα από ό,τι σε άλλους τομείς. Αλλά τι γίνεται για παράδειγμα, στον τομέα, ε, στο κεφάλαιο 1α, στο τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Γιατί εκεί πέρα υπάρχει κίνδυνος να μην μαζέψουμε και να μην καταφέρουμε να ορίσουμε ποσά. Άρα το θέμα που θα πρέπει να συζητήσουν οι ομάδες, θα πρέπει να συζητήσει και η ομάδα εργασίας, κάποια στιγμή θα πρέπει να το αποφασίσουμε. Εγώ μόνο τη δική μου άποψη σας παρουσίασα. Για μας είναι εύκολο αυτό, αλλά μπορεί αυτό να προκαλέσει διάλυση του Κοινοβουλίου κάποια στιγμή για κάποιους τομείς. Το θέμα των ποσών μπορεί να καταστήσει το Κοινοβούλιο σε κάποιες περιπτώσεις αδύναμο εταίρος στις διαπραγματεύσεις. Ένα άλλο παράδειγμα και θα μας... Ε, ξέρουμε όλοι πώς έχει κατάσταση στο Συμβούλιο, πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη πλειοψηφία χωρών οι οποίοι ζητούν ε, σωστή χρηματοδότηση του τομέα συνοχής. Άλλα ε, κράτη λένε ότι το 1% είναι πολύ υψηλό ποσοστό. Το Κοινοβούλιο είχε πει 2013 5% είναι κάτι το οποίο χρειαζόμαστε προκειμένου να χρηματοδοτούνται οι στόχοι της στρατηγικής της Λισαβόνα. Αλλά αν δεν θέλουν τα κράτη-μέλη αυτή την ε, χρηματοδότηση θα πρέπει τα κράτη-μέλη να διευκρινίσουν ποιες προτεραιότητες έχουν. Ποιες προτεραιότητες θέλουν να αφαιρεθούν από τη λίστα, καθότι δεν είναι πλέον χρηματοδοτήσιμες. Θέλουν την ε, αναπτυξιακή πολιτική, την έρευνα και την ανάπτυξη. Να σας αναφέρω δύο μόνο παραδείγματα ενδεικτικά. Και παράλληλα θα πρέπει να έχουν υπόψη και στις περαιτέρω διεργασίες τους και αυτό ενδεχομένως ε, να μας ε, οδηγούσε, αν θέλετε, και στις κόκκινες γραμμές μας σε μια δύσκολη κατάσταση. Αν το, αν το Συμβούλιο δεν μας υποβάλλει μια σωστή πρόταση, χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες για τις μεμονωμένες κατηγορίες, και αν το Κοινοβούλιο αναγκαζόταν να αποφανθεί αρνητικά θα χρειαζόμασταν και το 2% το οποίο αμφισβητείται από πολλά κράτη-μέλη. Αυτό για μένα δεν θα αποτελούσε κρίση, κυρίες και κύριοι, γιατί θα συνεχίζαμε να δουλεύουμε με βάση κάποια αριθμητικά στοιχεία, κάποια νούμερα. Απλά το θέτω αυτό ως σκέψη, να το συνειδητοποιήσουμε όλοι ως κοινοβούλιο τι θα είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε και τι όχι, γιατί θα είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε και γιατί όχι γιατί κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ποια θα είναι η πρόταση της Δανικής Προεδρίας τον Ιούνιο. Θα πρέπει οι ομάδες να αποφασίσουν η καθεμία από μόνη της ποιο οδό προτίθεται η καθεμία να ακολουθήσει. Και οι εθνικές κυβερνήσεις να πούν ότι εντάξει θα συνεχίσουμε επί αυτής της βάσης. Και επίσης είναι σαφές ότι όσο πιο δύσκολα είναι τα ποσά, τόσο πιο μεγάλη ευελιξία θα πρέπει να δείξει το Κοινοβούλιο, γιατί η εμπειρία με τις δύσκολες αυτές διαπραγματεύσεις κατά το παρελθόν μας δείχνει ότι χρειάζεται περιθώριο ελιγμού σε αυτές τις περιπτώσεις και αυτό προβλέπεται και στην έκθεση Γκαρίγκα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά θα προσπαθήσουμε την Τετάρτη να παρουσιάζουμε και να διευκρινίσουμε την Τετάρτη στην ομάδα εργασίας. Και νομίζω ότι θα, θα συζητήσει αυτά και η διάσκεψη των Προέδρων. Και όλα αυτά που είναι αφιλεγόμενα νομίζω ότι μπορούμε να τα επιλύσουμε στην πάρδο της εβδομάδας. Θέλετε να προσθέσετε κάτι. Να προσθέσω κάτι σύντομα σε αυτά που είπε ο Ρέινερ. Συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπε για την ανάγκη να συντονίσουμε τις θέσεις μας για τη συνολική στρατηγική. Ε, μπορούμε να παίξουμε ρόλο μόνο αν έχουμε ενιαία θέση. Δηλαδή, ουσιαστικά ε, το Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια και οι διάφορες πολιτικές ομάδες να δουν τι άποψη θα έχουν. Αλλά και εμείς ως σημαντική επιτροπή, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, θα πρέπει να βοηθήσουμε στην επίτευξη αυτής της ενιαίας θέσης. Η Δανέζικη Προεδρία θα ξέρετε ότι διενεργεί τις πρώτες συνεδριάσεις και συζητάει διάφορα θέματα που αφορούν το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Τα θέματα της περιφερειακής ανάπτυξης κατά πάσα πιθανότητα θα συζητηθούν στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων τον Απρίλιο. Ε, εν ώψη αυτού του Συμβουλίου, η Δανέζικη Προεδρία θέτει ερωτήσεις και περιμένει απαντήσεις από τα κράτη-μέλη. Και γιατί σας το λέω αυτό. Αυτό συνδέεται με την συζήτηση για τα αριθμητικά στοιχεία. Όταν η Δανέζικη Προεδρία έβαλε συζήτηση τα νούμερα, υπήρχαν τρεις ομάδες χωρών. Κάποιες χώρες που είπαν «Μ' αρέσει η πρόταση της Κομισιόν», κάποιες άλλες χώρες που είπαν ότι είναι πολύ νωρί για να συζητήσουμε τα αριθμητικά στοιχεία και η τρίτη ομάδα χωρών που ήθελαν σαφή μείωση των αριθμητικών στοιχείων. Υπήρχε και μια άλλη ομάδα χωρών, η Απούσα, και που ήθελαν ε, υψηλότερα αριθμητικά στοιχεία. Νομίζω ότι θα πρέπει να, εμείς να επικοινωνήσουμε καλύτερα με τα εθνικά κοινοβούλια. Σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γίνεται μια διάσκεψη κοινή μεταξύ του δικού μας Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και υπάρχει σήμερα το απόγευμα ένα σημείο προσυζήτηση ε, για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. 21 και 22 Μαρτίου το Κοινοβούλιο οργανώνει μία διάσκεψη ακριβώς για το ίδιο θέμα, για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, με τη, συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων και των Κυβερνήσεων. Θα ήθελα να έρθει σε επαφή με τα δικά σας κοινοβούλια, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Δύο-τρία σημαντικά θέματα ακόμα που πρέπει να συντηθούν για την πρόταση της Κομισιόν. Η πρόταση της Κομισιόν εστιάζει στο συνολικό πακέτο και στα συνολικά ποσά. Υπάρχουν όμως κάποιες αλλαγές και υπάρχουν πολλές, ε, πολλές αλλαγές στην ε, πολιτική συνοχής. Η Προεδρία ακριβώς αυτό το θέμα θέτει προς στα κράτη-μέλη. Και αυτό θα συζητήσει το Συμβούλιο ε, τον Απρίλιο. Το θέμα της αιρεσιμότητας θα πρέπει να συνδέεται με μακροοικονομικά στοιχεία ή όχι. Στην πρόταση της Κομισιόν Ε, οι κυρώσεις ε, που αναφέρονται στο ευρωπαϊκό εξάμεινο αφορούν μόνο την πολιτική συνοχή. Υπάρχει μια προσφυγή εναντίον της Ουγγαρίας τώρα. Στην τελευταία συνεδρίαση συζητήθηκε αυτό. Και η πολιτική συνοχή μπορεί να είναι πραγματικά ε, το θύμα αν συνεχίσουν τα πράγματα προ την ίδια Η συγχρηματοδότηση και η προχρηματοδότηση. Το θέμα της, ε, περιφερειακής, κάλυψη γεωγραφικής κάλυψης ε, των ταμείων. Ε, η κατανομή των περιφερειών, λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, μεταβα... περιοχές σε μετάβαση, απομακρυσμένες περιοχές, αεροκατοικημένες περιοχές. πώς αποφασίζει η Κομισιόν να κατανείμει τα 336 δι, Το ανώτατο όριο είναι αποδεκτό. Στην πρόταση της Κομισιόν υπάρχει αυτό το ανώτατο όριο του 12,5% ως προς τη δυνατότητα χρήσης των κονδυλίων των ταμείων. Ποια θα είναι τα κριτήρια κατανομής. Ε, περιφερειακός πλούτος, ε, απασχολησιμότητα ε, κτλ. Εδώ έχουμε διαφορετικές θέσεις ε, σε διαφορετικές χώρες. Ε, το Connecting Europe Facility. Ε, μεταφέρονται 10 δισεκατομμύρια από τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής εκεί, για αυτό το facility. Όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να συζητηθούν. Και νομίζω ότι εμείς στην, ε, στην Επιτροπή Ρέτζιο πρέπει να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Πρέπει να συζητήσουμε αυτά τα θέματα μαζί με... Και εμείς από την πλευρά μας όταν τα συζητάει και το Συμβούλιο Γενικά πρέπει να συζητήσουμε τη νέα οργάνωση της πολιτικής συνοχής. Συνάδελφοι, να σας ξεκαθαρίσω το εξής. Okay, ε, Και εμεί έχουμε προσκληθεί στην συνάντηση με τον πρόεδρο Σούλτ την Τετάρτη. Οπότε την... το Μάρτιο προτείνω να συζητήσουμε όλα τα σχετικά με το ε, πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και να αποφύγουμε τη συζήτηση αυτού του θέματος σήμερα γιατί δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Ίσως θα μπορούσαμε να δεχτούμε δύο-τρεις ερωτήσεις, αλλά μόνο ερωτήσεις παρακαλώ, προς τον εισηγητή, ε, προς τον εισηγητή της, ε, για τον προπολογισμό. Οπότε, Λαμπέρ, μόνο αν έχεις ερώτηση παρακαλώ, ζήτησε το λόγο. Ο ε, Ιαν Νίλσεν επίσης ζήτησε το λόγο. Μόνο ερωτήσεις όμως παρακαλώ. Πρόεδρε. Eh, Πρόεδρε, είστε πάρα πολύ αυστηροί σήμερα στο θέμα αυτό. Τι να κάνουμε, θα πρέπει να σας ακολουθήσουμε τις οδηγίες σας, αλλά... Μία ερώτηση να κάνω και δύο παρατηρήσεις. Καταρχάς, είναι πάρα πολύ καλό το ότι συνεννοούμαστε έτσι άμεσα, γιατί δεν είναι δυνατόν το Συμβούλιο να κινείται βαθμιαία και εμείς να περιμένουμε μέχρι τον Οκτώβριο. για να καταθέσουμε αυτή την ενδιάμεση πρόταση. Θα πρέπει να τηρήσουμε λοιπόν τα όσα αποφασίσαμε στην έκθεση Γκαρίγκα και το πράττουμε αυτό και στην Επιτροπή αυτή. Ε, ισχύουν όλα τα... Έχουμε συζητήσει όλες τις νέες αρχές για την πολιτική συνοχή. Με την έκθεση Πίπερ, για παράδειγμα, που αξιολόγησε την προηγούμενη φάση και έδωσε κατευθυντηρίες γραμμές για το μέλλον. Τα συζητήσαμε λοιπόν όλα αυτά μία φορά, άρα είμαστε έτοιμοι με τα τμήματα αυτά. Για να ακουστική η φωνή μας. Γιατί δικαίω αναφέρει, για παράδειγμα, ο συνεισηγητή. Κοιτάξτε, η γεωγραφική, για παράδειγμα, το γεωγραφικό εύρο. Κάποια πράγματα είναι απαράδεκτα για το Κοινοβούλιο. Δεν είναι δυνατόν η πολιτική συνοχή να περνάει στι νέε προοπτικέ του 2020 και αυτό να ισχύει παράλληλα για, μία, για ένα τμήμα μόνο τη γεωγραφική περιφερεια. Υπάρχουν ε, κάποια πράγματα που το Κοινοβούλιο μπορεί να απαντήσει μόνο αρνητικά. Μόνο αρνητικά. Αυτοί μπορούν να μας προτείνουν ό,τι θέλουν, αλλά κάποια πράγματα πολιτικώς πώς δεν είναι επιτρεπτά. Τα έχουμε συζητήσει λοιπόν ως Επιτροπή. Η ερώτησή μου τώρα για τα ποσά. Και οι δύο γνωρίζουμε την συστηματική ε, που ακολουθείτε σε ό,τι αφορά την συνοχή. Ατυχής. Ο τρόπος που αυτό μεταφράζεται στις διάφορες περιφέρειες αποτελεί ένα συνεκτικό σύνολο. Άρα δεν υπάρχει οποιαδήποτε ανάγκη να το διαλύσουμε αυτό το σύστημα. Μιλάμε για μικρές προσαρμογές. Αλλά άλλα πράγματα είναι στην δική σας αρμοδιότητα, για παράδειγμα για το κάπινγκ. Θα πρέπει να περάσουν και στην Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων, γιατί είναι πολύ ειδικά θέματα. Εμείς θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε με τα ποσά. Και θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια τον Σεπτέμβριο το τι επιθυμούμε. Ιδάλλως έχουμε την αίσθηση ότι μας ξεποπουλιάζουν. Προτού έχει φτάσει η στιγμή. Ελπίζω λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο να ενημερωνόμαστε μέσω των διάφορων ομάδων εργασίας. Uh, Μία ερώτηση και ένα σχόλιο. Ένα από τα πιο έντονα επιχειρήματα για μια νέα και μοντέρνα πολιτική συνοχής είναι ότι η πολιτική συνοχής εφαρμόζει και άλλες πολιτικές, όπως την πολιτική ε, για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, την πολιτική έρευνας και άλλες πολιτικές. Δεν είναι ισχυρό επιχείρημα αυτό όταν συζητάμε με τα εθνικά κοινοβούλια, με τις, με κυβερνήσεις, να το προτάξουμε για να τους πιέσουμε. Δεύτερον, και σύντομα, σε ό,τι αφορά τις ε, περιοχές στην Σουηδία και Φιλανδία, πρέπει να πούμε από πλευράς Κοινοβουλίου ότι αναγνωρίζουμε την ιδιαιτερότητα αυτών των ε, περιοχών με βάση τη συνθήκη. Αυτό πρέπει να το πούμε στο έγγραφό μας. Ε, Ερικα Μάνερ, τελευταία ερώτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να τονίσω μερικά σημεία. Μας απογοητεύει το γεγονός ότι δεν έχουμε ακριβώς τα επαρκή αριθμητικά στοιχεία, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε αποφάσεις. Γι' αυτό ακριβώς θα ήθελα να μου πείτε αν θα λάβετε πιο σαφείς πληροφορίες από πλευράς Επιτροπής. Δεύτερον, θα ήθελα να μου δοθούν πληροφορίες για τις υποχρεώσεις. Θέλω να δω τι θα γίνει με τις πιστώσεις υποχρεώσεων. Τι θα γίνει με τις δεσμεύσεις υποχρεώσεων. Συμφωνώ με τον κύριο Νίλσεν που μίλησε για τις ε, απομακρυσμένες περιοχές, τις ε, αεροκατοικημένες περιοχές. Τι ποσά θα τους δοθούν. Ε, τα ποσά αυτά που τους δίνονται είναι μικρότερα. Αν τα νούμερα αυτά που μας παρουσίασε η Κομισιόν είναι σωστά, τότε σημαίνει ότι υπάρχουν σοβαρότατες περικοπές των πιστώσεων για αυτές τις περιοχές. Σας ευχαριστώ για τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Δεν ξέρετε ποιοι είναι οι εσωτερικοί μας κανόνες. Ε, η Επιτροπή ε, Προϋπολογισμών μιλάει για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και για τις, τα έσοδα και τα έξοδα. Εσείς, εσείς μιλάτε ε, και γνωμοδοτείτε για την πολιτική συνοχής. Και όπου μπορούμε θα σας υποστηρίξουμε. Αλλά δεν μπορούμε να παρέμβουμε σε αυτά τα λεπτομερή θέματα. Αυτά είναι δικά σας θέματα. Πρέπει να μιλήσουμε λοιπόν για το περιεχόμενο με τρόπο ούτω ώστε αυτή η προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω που δεν χρησιμοποιήθηκε επί Πολωνικής Προεδρίας αλλά που χρησιμοποιείται τώρα επί Δανικής Προεδρίας να μην γίνει αυτόματα αποδεκτή. επανέρχομαι σε αυτή την πολιτική συμφωνία του 2005 που λέει ότι το Κοινοβούλιο θα μιλήσει για τα δικά του προγράμματα και θα ε, ολοκληρώσει την πρώτη ανάγνωση. Το Συμβούλιο θα φτάσει σε μερική συμφωνία για την πρόταση χωρίς τα νούμερα και τα άρθρα που αφορούν τις ε, δημοσιονομικές διατάξεις. Και τρίτον, τα δύο θεσμικά όργανα με βάση τις θέσεις τους θα αρχίσουν Προκαταρτικέ προτάσεις για την νομοθετική πρόταση με την εξέταση των άρθρων που αφορούν ε, τη δήλωση για τον προπολογισμό, τον προπολογισμό ούτω ώστε να φτάσουν σε κοινή θέση. Και αφού συμφωνήσουν επί του προσχεδίου θα μιλήσουν και για τα νούμερα ούτω ώστε να συμφωνήσουν ε, και επί των 70 ε, προγραμμάτων όπου υπάρχει συναπόφαση. Αυτή ήταν η συμφωνία αυτό είχαμε συμφωνήσει, ούτω ώστε να αποφύγουμε αυτή την ε, λήψη αποφάσεων από πάνω προς τα κάτω. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξουμε τη μέθοδο εργασίας. Και να πούμε στο Συμβούλιο, εμείς ετοιμάζουμε την πρώτη ανάγνωση, Συμβούλιο. Σταματάμε και μετά ετοιμάζουμε και κάνουμε ε, προκαταρ... προκαταρτικές συζητήσεις. Αυτό το κείμενο μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε τις διαπραγματεύσεις πριν φτάσουμε στο πραγματικό νούμερο του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και τι σημαίνει αυτό για την πολιτική συνοχή, για σημαίνει για την έρευνα κτλ. Δεν χρειάζεται κάθε μέρα να μιλάμε για νούμερα όλοι. Ξέρουμε το γενικό πλαίσιο της έκθεσης Γκαρίγκα. Ξέρουμε ποιο είναι, ποια είναι η θέση της Κομισιόν που είναι χαμηλότερη. Ξέρουμε ποια είναι η θέση στο Συμβούλιο. Δεν υπάρχει ομοφωνία, σε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Δεν υπάρχει περίπτωση να ακολουθήσει αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο ή την Κομισιόν. Αυτή είναι η πολιτική πραγματικότητα. Αλλά για να του πείσουμε θα πρέπει να του πούμε. Πρέπει να συζητήσουμε για τα θέματα σύγκληση. Πρέπει να συζητήσουμε τι νέε κατηγορίε. Πρέπει να συζητήσουμε όλα τα άλλα στοιχεία που ανέφερε ο κύριο Νίλσεν και ο κύριο Φανίστελ Ρόι. Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την πολιτική συμφωνία. αν την πετύχουμε βέβαια ή θα συμπεριλαμβάνονται μάλλον. Και αυτό θα ενισχύσει το, τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό. Στη Διαθεσμική Συμφωνία υπάρχει μια περιγραφή του πλαισίου, όπως είδατε, και μια δυνατότητα για συμφωνίες. Δεν μπορούμε στις διαπραγματεύσεις να συζητήσουμε τα πάντα. Ε, όλα αυτά που δεν πετύχαμε στην νομοθετική διαδικασία δεν μπορούμε να τα ξανασυζητήσουμε. Μην, ξεχνάτε την συζήτηση για την ιδιωτική χρηματοδότηση. Αυτό συμπεριλήφθηκε συνεχεία στη διαθεσμική συμφωνία ε, εκ των υστέρων ως δυνατότητα. Ε, και με αυτόν τον τρόπο απορροφούμε λεφτά από την πολιτική συνοχή που αλλιώς θα μπορούσαμε να απορροφήσουμε. δεν μπορούμε να παρεμβαίνουμε σε κάθε φάση της νομοθετικής διαδικασίας. Θα τους πούμε, εμείς περιμένουμε και θα παρέμβουμε την κατάλληλη στιγμή. Είμαστε έτοιμοι να σας πλαισιώσουμε. Αν μπορούμε να συμφωνήσουμε επί μια τέτοια δήλωση, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για τι επιτροπέ, ούτω ώστε να αναγκάσουμε το Συμβούλιο να κάνει κάποιε προ... προκαταρκτικέ συζητήσει για να δούμε πού βρισκόμαστε στο τέλο τη πρώτη ανάγνωση χωρί να έχουμε και την τελική, την ψηφοφορία. Γιατί πώ θα ψηφίσουμε χωρί νούμερα, αλλά να, να προετοιμάσουμε όλα τα υπόλοιπα, ούτω ώστε να έχουμε μια πραγματική θέση για διαπραγμάτευση. Σε περίπτωση που υπάρχουν προβλήματα στο Συμβούλιο, να δείξουμε ότι εμεί τουλάχιστον είμαστε έτοιμοι ε, να πετύχουμε αποτελέσματα και ούτω ή άλλω περιμένουν κάτι τέτοιο οι περιφέρειε. Uh, Δύο λόγια μόνο. Είναι σαφή τα πράγματα με τα αριθμητικά στοιχεία. Έχουμε την πρόταση Κομισιόν. Σα υπενθυμίζω ότι 354 εκατομμύρια είναι για τα 7 χρόνια το δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Κομισιόν προτείνει 336, δηλαδή 20 δισεκατομμύρια λιγότερο σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο 2007-2013. Και μετά ε, γίνεται κατανομή, αναπεριφέρεια, περιφερειακά ταμεία ανάμεσα σε, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 και των 12 κλπ. Όλα αυτά τα στοιχεία τα έχουμε. Αλλά ό,τι και να πούμε δεν είναι αρκετό. Η θέση του Κοινοβουλίου ήταν 385 δισεκατομμύρια τουλάχιστον. Πολύ περισσότερο δηλαδή από αυτό που προτείνεται, τα 336. Οπότε φαντάζομαι ότι διατηρούμε τη θέση μας. Αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα που πρέπει να συζητήσουμε συμπεριλαμβανομένου και αυτού που είπατε. Η Κομισιόν προτείνει ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο για να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα όλων των ταμείων μαζί. Ε, επίσης, ε, να υπογραφούν ε, συμφωνίες εταιρική σχέση με τις, ε, τα κράτη-μέλη, να εξετάσουμε το, τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων ταμείων κλπ. Όλα αυτά είναι συζητήσιμα και χωρίς να μιλήσουμε για τα νούμερα. Θα μιλήσουμε για τα νούμερα, αλλά εστιαστούμε σε πρώτα σε αυτά τα θέματα. Ε, πρόεδρος, να προσθέσω το εξής. Ε, μια πρόσθετη επιπλοκή προκύπτει από το, το γεγονός ότι με τη συναπόφαση αποφασίζεται το, ε, το ρυθμιστικό πλαίσιο. Και πολλά πράγματα τα πήρε το Συμβούλιο από το ρυθμιστικό πλαίσιο και τα μετέφερε στην ομάδα αυτών που θα αποφασίσουν για τον προϋπολογισμό. Κάτι που από νομικής πλευράς είναι αμφισβητήσιμης ε, ορθότητας. Γιατί αυτοί θα εξετάσουν βέβαια τις οικονομικές, τα, οικονομικά στοιχεία, αλλά θα επηρεάσουν με αυτόν τον τρόπο πάρα πολύ τη δική μας δουλειά. Συνεπώ θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να μην επιτρέψουμε στο Συμβούλιο μέσω διαφορετικής οδού να αποφασίσει το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Ναι, και κάτι ακόμα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμεί χαιρόμαστε που οι Υπουργοί Οικονομικών δεν αποφασίζουν τον προπολογισμό. Από τη δική μα πλευρά αυτό είναι καλό. Γιατί αν τα αποφασίζαν αυτοί θα είχαν πολύ χαμηλό προπολογισμό. Ε, είναι σημαντικό αυτό να αποφασιστεί από το ε, Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και ε, το ΕΚΟΦΗΝ θα ενημερώνεται αλλά η απόφαση θα ληφθεί από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Βέβαια, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων δεν μπορεί να αναλάβει τι αρμοδιότητε των άλλων συμβουλίων. Οπότε εδώ μιλάμε για περιφερειακή πολιτική, Συνεπώ ε, αυτή θα πρέπει να συζητηθεί και αλλού, όχι μόνο στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Πάντω θα πρέπει να είμαστε πολύ αποφασιστικοί ενώπιον εναντί του, του Συμβουλίου. Εμεί μιλάμε με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ωραία, να κλείσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ κύριε ε, Μπέγκε που ήρθατε εδώ και τους δυο σας. Ε, ελπίζω θα ξανασυζητήσουμε το θέμα αυτό. Άντριου. Ναι, ναι, σωστά, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και το συγγητέ. Κύριε Μπέγκε, μια ερώτηση. Πότε μπορούμε να αναμένουμε την ε, απόφαση Επιτροπής Προπολογισμού για την ενδιάμεση έκθεση τον Οκτώβριο, είπατε ενδεχομένω. Για το ψήφισμα και την ενδιάμεση έκδοση, εγώ σας μίλησα για μια πρόταση των εισηγητών. Η ομάδα επαφής θα τη δει την Τετάρτη και θα περάσει στην διάσκεψη των Πρόεδρων. Μετά, αφού ληφθούν αυτές οι αποφάσεις, θα προετοιμάσουμε το χρονοδιάγραμμα κάτι που θα, μας, θα, δώσει, αρκετό χρόνο στις επιτροπές να προετοιμάσουν την γνωμοδότησή τους. Πρόκειται λοιπόν για ενδιάμεση έκθεση που θα είναι έτοιμη στις αρχές Οκτωβρίου. Το, για το Μάιο θα προετοιμάσουμε ένα ψήφισμα ε, με κατευθυντήρες γραμμές ή κόκκινες γραμμές αν θέλετε για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου. Όμω η ενδιάμεση έκθεση θα, μπει πιο, ε, θα εξετάσει πιο λεπτομερώς τα πράγματα από ότι ένα ψήφισμα. Το ψήφισμα θα αντικατοπτρίζει απλώ τη γενική θέση του Κοινοβουλίου και θα δίνει γενικέ κατευθυντήρε γραμμέ για το τι έχει να πει το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ωραία. Α περάσουμε στο επόμενο σημείο τη ημερησία διάταξη με τεράστια καθυστέρηση. Γνώμη του Ελεκτικού Συνεδρίου. Είναι εδώ ο κ. Φαζάκα. Ε, το, ε, το Ελεκτικό Συνέδριο έχει προετοιμάσει επίση και την αξιολόγηση του ρυθμιστικού πλαισίου για, την, για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο κ. Ε, Φαζάκας είναι εδώ να μας, την, ε, να μας παρουσιάσει αυτή την ε, γνωμοδότηση. Πρόεδρε, αγαπητή Τανούτα, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη μοναδική αυτή τη ευκαιρία να παρουσιάσω την άποψη του ελεκτικού συνεδρίου σχετικά με τις κοινέ διατάξεις για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία για την, περίοδο αυτή 2014-2020. Είναι μεγάλη τιμή που έχω την ε, ευκαιρία να συζητήσω την, με την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι η καθήλυνα αρμόδια Επιτροπή του Κοινοβουλίου. Πρωτού περάσω σε λεπτομέρειες, θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Κωνσταντσε Αγγελά Κρέιλ και τον κύριο Λάμπερτ Φανίστε Ρόι, που είναι οι εισηγητέ για την υψηλή ποιότητα του εγγράφου εργασίας. Με, πραγματικά με ενθάρρυνε πάρα πολύ το γεγονός ότι ακολουθείται μια κοινή προσέγγιση και μάλιστα ο τρόπος εργασία σας ε, συμπληρώνει το δικό μας. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω καταρχάς ότι το σχέδιο ε, νομοθεσία σε την περίοδο 2014 έως 2020 θέτει και κάποια πολιτικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να είναι αρμοδιότητα πολιτικών. Ημών δηλαδή των ε, δημοκρατικά εκλεγμένων εκπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν αποφύγαμε να υποστηρίξουμε ή να καταδικάσουμε οποιαδήποτε πρόταση του κανονισμού γιατί από εσάς, από τους νομοθέτες εξαρτάται κατά πόσον θα συμπεριλάβετε και θα δεχτείτε τις προτάσεις αυτές ή όχι. Το ελεκτικό συνέδριο θεωρεί ότι ρόλος του είναι να να παρέχει καθοδήγηση σε σχέση με αυτά που προτείνονται με τις δικές του συστάσεις και τα δικά του πορίσματα μετά από τις θετικές εμπειρίες με την γνωμοδότησή μας από το 2005 σε ό,τι αφορά τον κανονισμό και την τρέχουσα περίοδο. Η γνώμη μας και η γνωμοδότησή μας βασίζεται σε κάποιες βασικές, ε, σε κάποια βασικά αποτελέσματα, απορίσματα των ε, πρόσφατων ελέγχων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα μέσα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, οι δράσεις που έχουν ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βελτιωθούν θέματα αποδοτικότητα στα κράτη-μέλη, ε, τα... και τα πορίσματα από την περίοδο του 2006. Παρουσιάζοντας την γνωμοδότηση αυτή, θα ήθελα να κοιτάξουμε παράγραφο παράγραφο τα πορίσματά μας. Πολύ φοβάμαι όμως ότι δεν έχουμε το χρόνο να το πράξουμε αυτό. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα τέσσερα πολύ σημαντικά στοιχεία να σας επισημάνω. Καταρχάς, η ίδρυση, η θέσπιση ενός νομοθετικού πλαισίου για τις δαπάνες σε θέματα συνοχής για την περίοδο 2014 2020 μας δίνει μια ευκαιρία να διευκρινίσουμε την προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία, θέτοντας προτεραιότητες. Προκειμένου να πετύχουμε λοιπόν αυτή την υπεραξία, το ελεκτικό συνέδριο προτείνει να κοιτάξουμε τα αποδεκτά αποτελέσματα με ε, κάποια κριτήρια αντικειμενικά. Ωστόσο, Παρά τη σαφή επικέντρωση στα αποτελέσματα, το προτινόμενο πλαίσιο για το 2014-2006 ουσιαστικά παραμένει ένα σύστημα βάσης του input, βάση και κινούμαστε μάλλον πιο πολύ προς την κατεύθυνση της συμμόρφωσης παρά προς την κατεύθυνση των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, ε, οι πόροι μπορούν να δαπανηθούν σε πάρα πολύ μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων και είναι πολύ περιορισμένη λοιπόν η απτή, το απτό αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής ε, ε, δράσης. Ε, η, κατά δεύτερον, η εξάντε αιρεσιμότητα αποτελεί ένα σημαντικό, μια σημαντική εξέλιξη. Από την άποψη αυτή και δεδομένων της σημασίας των πόρων C SF είναι πολύ σημαντικός ο τομέας αυτός. Κατά τρίτον, διάφοροι εμπειρογνώμονε, ε, ανα, μάλλον διαφορετικά σημεία εμπειρογνωμοσύνης αναβάλλονται για ένα μετέπειτα χρονικό στιγμίο, σημείο. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά με, το, με τις πράξεις εξουσιοδότηση, εξουσιοδότηση και τις ελευθερικές πράξεις. Οι πράξεις κατά εξουσιοδότηση όμως υποτίθεται ότι είναι μη ουσιώδη στοιχεία της ευρωπαϊκή νομοθεσία. και όμω εδώ πραγματεύονται πολύ ουσιώδη στοιχεία τη πολιτική συνοχή και μπορεί να περνούν και πέρα από συγκεκριμένα στοιχεία και να έχουν επιπτώσεις και για άλλες νομοθεσίες. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει συνοχή μεταξύ των διαφόρων αυτών τομέων και στον όλο κανονισμό συνολικά. Επίσης είναι σημαντικό να τονίσουμε την αναγκαιότητα να υπάρχει συμμόρφωση μεταξύ του κανονισμού κοινών διατάξεων και, τον, και του δημοσιονομικού κανονισμού. Τέταρτο σημείο. Η προτινόμενη μείωση των ανώτατων ποσών για εθνικές πολιτικής και η μακρονομική ρεσιμότητα θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο εντελεχούς ε, μελέτης για να μην έχουν αρνητικές επιπτώσεις. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να αναλύσουμε τα αίτια ε, περιορισμένων δαπανών γιατί αν θέλετε η περιορισμένη απορρόφηση κάποιων περιοχών ε, οφείλεται κυρίως σε περιορισμένες διοικητικές ε, ικανότητες και άρα αυτή η μείωση των ανώτατων ορίων μπορεί να θεωρηθεί περιοριστικό μέτρο, το οποίο θα, θα ε, επηρεάσει ιδιαίτερα τις πιο ευάλωτες περιοχές και δεν μας δίνει ουσιαστικά στοιχεία για την δυνατότητα απορρόφησης και για το επίπεδο ανάπτυξης. Και η γενική μείωση αυτών των ανώτατων ορίων μπορεί να επηρεάσει και περιοχές με υψηλό ποσοστό ανάπτυξης τα επιτεύγματα τώρα το, της ε, μακροοικονομικής απόδοσης ε, αποτελούν κάτι το οποίο ωφελεί όλα τα κράτη-μέλη. Η προτινόμενη μακροοικονομική αιρεσιμότητα έχει ως σκοπό να διευκολύνει ακριβώς την πρακτική εφαρμογή των μέτρων αυτών. Αλλά αυτό θα προαπαιτήσει μια εντελεχή ανάλυση των συγκεκριμένων έμεσων και άμεσων επιπτώσεων και σε επίπεδο κρατών μελών και σε επίπεδο περιφερειών. Η αυξανόμενη, αν θέλετε, διακοπή προγραμμάτων σε, περιφερειακά, σε περιφερειακό επίπεδο μπορεί να διακινδυνεύσει την επίτευξη κοινά αποδεκτών στόχων. Και μπορεί να επηρεάσει και τον, ε, την ε, τα, τα, τα αποτελεσματικά συστήματα ελέγχου. Δεν θα συνδράμει ούτε στη μακροοικονομική σταθερότητα στην, ε, στο κράτος, ούτε στη συγκεκριμένη περιφέρεια. Να σας επιθυμίσω ότι το ελεκτικό συνέδριο ήταν εκείνο που πάντα ζητούσε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναστέλνει ε, άμεσα ε, τέτοιους πόρους συνοχής σε περίπτωση ατασταλιών. Αλλά αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η μακροοικονομική αιρεσιμότητα, περνάει σε άλλο επίπεδο. Δεν θα πρέπει να τα συγχαίουμε αυτά. Ξέρετε ότι πολλές φορές αυτά μπορεί να, να φανούν αντιπαραγωγικά. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κάτι το οποίο μπορεί να αναστείλει τη δημιουργία θέσεων εργασίας ο κανονισμός μπορεί να διακινδυνεύσει πολιετή προγράμματα σε περιφερειακό επίπεδο και μπορεί να δημιουργήσει ένα φαινόμενο χιονοστιβάδας, ε, επηρεάζοντα πολλές συμβάσεις σε διάφορες εταιρείες από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και η διακοπή χρηματοδότηση τέτοιων τοπικών έργων βάσει μακροοικονομικών παραγόντων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές νομικές αβεβαιότητες και σε νομικά προβλήματα. Τώρα, τώρα σε ό,τι αφορά την ε, διαχείριση τώρα που ε, με έχουν καλέσει στην κομπού την Τετάρτη, θα έχω την ευκαιρία, θεωρώ, να συνεχίσω τα τέσσερα αυτά σημεία σε λεπτομέρεια και νομίζω ότι καλύτερο θα ήταν να λάβατε τα σχετικά πορίσματα από τον κύριο Ντέρεκ. Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι θεωρώ τα πορίσματα του εγγράφου εργασίας σας και της γνωμοδότησης του ελεγκτικού συνεδρίου υποστηρίζουν το ένα το άλλο. Ελπίζω ότι οι δείκτες σας θα ληφθούν υπόψη στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα αποτυπωθούν ανάλογα και στον τελικό κανονισμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι έχουν να θέσουν διαφημιστικά ερωτήματα. Νομίζω ότι η θέση σας είναι σαφής. Μερικές φορές μας εκπλήττει κιόλα, διότι σε πολλές φορές, πολλές φορές <laughs> οι συζητήσεις με το Ελληνικό συνέδριο είναι πολύ πιο ε, ε, αυτή τη φορά εκφράζεται πιο πολύ τις δικές μας απόψεις. <laughs> Καλή καλή κατάσταση αυτή. Ε, Λαμπέρ, έχεις ε, κάποια ερώτηση. Ε, Στην Επιτροπή αυτή, Πρόεδρε, πάντα προσπαθούμε να βρούμε τρόπους συνεργασίας και είναι πάρα πολύ καλό το ότι υπάρχει ανταπόκριση. Θα ήθελα να σας θέσω το θέμα του κάπινγκ και της ε, όλης λογικής πίσω από αυτό ότι μπορεί τα αποτελέσματα να είναι πολύ διαφορετικά από ότι είναι η πρόθεση της πολιτικής συνοχής. Αυτά μας τα αναφέρατε και εγγράφος. Γιατί και για μας είναι σημαντικό στη συζήτηση που θα διεξαχθεί τώρα. Υπάρχει η σκέψη λοιπόν και σε μας ότι υπάρχει μια ανισορροπία όχι μόνο από πολιτικής άποψης αλλά και από πλευράς περιεχομένου. Θα θέλαμε να μας παρουσιάσετε ε, τους λόγους που σας οδήγησαν στα πορίσματα αυτά για θέματα μακροερεσιμότητας Δεν έχουμε την εντύπωση ότι αυτά τα θέματα μακροπρόθεσμης αιρεσιμότητας τίθενται μόνο εδώ. Έχουμε την εντύπωση ότι προέρχονται από πολύ πιο πάνω από το Six από συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα λαθεσμικά όργανα. Και εδώ θα ήθελα να μας παρουσιάσετε τους λόγους που σας οδήγησαν στα πορίσματα αυτά, αλλά διαπιστώνω ότι συγκλίνουν οι απόψεις μας. Και πραγματικά μας είναι πολύ χρήσιμα τα στοιχεία που μας παρουσιάσατε. Αναζητώ μία μέθοδο προκειμένου στην φάση των τροπολογιών να μπορούμε να έχουμε και επαφή μαζί σας. Γιατί όπως ξέρετε ο διάβολος στις λεπτομέρειες κρύβεται. Προκειμένου να υπάρχει μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας. Σας ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ για τα στοιχεία που μας παρουσιάσατε. Το ε, Ελεκτικό συνέδριο η ε, και μάλιστα κάποιε λεπτομέρειες που εκεί βρίσκεται ο διάβολο πάντοτε. Ο συνάδελφος, όπως είπε ο συνάδελφος από το Ελεκτικό συνέδριο, ε, είμαι υπεύθυνο για την ομοδότηση της ε, Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού. αν θέλετε μπορείτε να την Διαβάστε πριν την ε, πέμπτη που θα συζητηθεί, αν, ε, αν έχετε αϊπνία. Αν δεν θέλετε να διαβάσετε όμως, να σας πω τρία-τέσσερα πράγματα που έχουμε συμπεριλάβει στην γνωμοδότησή μας. Πρώτον, η πρόβλεψη για τα ποσοστά λάθους που γίνεται ετησίως. Συνήθως είναι 5 με 7%. Ε, δεν περνάμε πάντοτε το μήνυμα μας ότι μιλούμε για λάθη και όχι για απάτη. Δεύτερον, δεν είμαι σίγουρος ότι αστιαζόμαστε στο σωστό θέμα, διότι αυτό το ποσοστό δεν μας λέει τίποτα για την αποτελεσματική χρήση των ποσών των κοντιλίων. Δεύτερον, ε, η μετάβαση σε ένα σύστημα που θα βασίζεται πιο πολύ στις ε, εξόδους παρά στις εισόδους. Στο output και όχι στο input. Και αυτό πρέπει να το σκεφτούμε για το μέλλον. Τρίτον, γίνεται η πρόταση από την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού να ε, κάνουμε περισσότερη διαπίστευση στο πλαίσιο των συστημάτων διαχείρισης, έτσι ώστε οι διαδικασίες των κρατών μελών να εγκρίνονται εκ των προτέρων από την Κομισιόν. Απ' την άλλη μεριά θα πρέπει να διασφαλίσουμε και ότι η ευθύνη για τη χρήση των κονδυλίων της συνοχής είναι ανοίξει την Κομισιόν. Θα πρέπει λοιπόν να αυτή η ισορροπία. Ένα άλλο θέμα είναι η απλούστευση. Μιλάμε συνεχώς γι' αυτό. Αλλά θα πρέπει να δούμε αν πρόκειται για απλοποίηση για τους δικαιούχους, για τα κράτη-μέλη, για τις περιφέρειες. Και εκτός αυτού να το υλοποιήσουμε κιόλας, γιατί πολλά, μιλάμε για το θέμα αυτό, αλλά δεν έχουμε κάνει και πολλά μέχρι τώρα. Η απλοποίηση θα πρέπει να εξασφαλιστεί. Χαίρομαι που το ελεγκτικό συνέδριο αμφισβητεί την ανάγκη μακροοικονομικής αιρεσιμότητας. Έτσι κι αλλιώς αυτή η πρόταση δεν έχει πολλούς φίλους πουθενά. Δεν καταλαβαίνω γιατί η Κομισιόν επιμένει. Επίσης υπάρχει το θέμα των αναστολών και των διακοπών. Το συζητούμε συχνά στην Επιτροπή μας. Το ερώτημα είναι αν, αν γίνονται αυτόματα οι αναστολές ή αν θα πρέπει να γίνονται συστηματικά. Δηλαδή, πριν γίνει οποιαδήποτε διακοπή ή αναστολή, να έχουμε περάσει προς συγκεκριμένα στάδια. Τέλος, μιλούμε για τα νέα χρηματοδοτικά μέσα, τα οποία θα είναι πολύ σημαντικά για μας, γιατί η πολιτική συνοχής ε, περικόπτεται από πολλές πλευρές, ε, οπότε οι περιφέρειες θα αναζητούν χρηματοδοτικά μέσα, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια ισορροπία, να έχουμε κανόνες για αυτά τα νέα χρηματοδοτικά μέσα και ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνονται εκταμιεύσεις ελαστικά, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες να αποφασίζουν τα ίδια και οι ίδιες ε, πού θα δαπανηθούν τα διάφορα ποσά. Πολλά λοιπόν καλύπτουμε στην έκθεσή μας που θα υποβάλω στην Επιτροπή ε, Ελέγχου του Προπολογισμού και κάποια στιγμή θα φτάσει και στα χέρια σας. Ευχαριστώ. Κύριος Ντόιτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγα... Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να πω το εξής καταρχήν. Καταρχά, το κείμενό σας είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο, πολύτιμο και τεχνικό. Και τίθενται μια σειρά από ερωτήματα στην έκθεση αυτή. Εγώ θέλω να σταθώ σε λίγα μόνο από αυτά τα θέματα, σε λίγα από αυτά τα ερωτήματα. Σε ποια φάση είμαστε τώρα. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολούμαστε με την περίοδο μέχρι το 2013 και δουλεύουμε επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας. Αλλά βέβαια θα μου πείτε ότι όλα είναι αλεξαρτημένα. Το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι ένα πακέτο. Έχουμε διάφορα κείμενα, διάφορα σχέδια κειμένων, τα οποία είναι υποσυζήτηση. Γι' αυτό ακριβώς το κείμενο του Ελληνικού Συνεδρίου είναι πολύ σημαντικό. Για να μελετήσουμε αυτό το κείμενο, θα πρέπει παράλληλα να μην ξεχνάμε την απόφαση που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα. Δηλαδή μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ουγγαρία εν προκειμένου, στα πλαίσια του, της διαδικασίας του υπερβολικού χρέους θα υποστεί κυρώσεις που αποφασίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι κυρώσεις αυτές βαραίνουν πολύ. Δηλαδή, αν το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ συμφωνήσει με την πρόταση της Επιτροπής, από το 2013 οι πόροι που θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει η Ουγγαρία θα μειωθούν κατά 29%. Τουλάχιστον αυτή είναι η πρόταση. Η βάση της πρότασης της Κομισιόν είναι ότι έκανε κάποιες προσωμιώσεις για το μέλλον. Από το 2004 η Ουγγαρία βρίσκεται στη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος. Και μάλιστα το 2011 και 2012 θα έχει ελλείμματα που δεν είναι τόσο υψηλά. Θα είναι κάτω του 3% λέει ο μιλητής. Ίσως όμως μετά το 2012 αυξηθεί αυτό το έλλειμμα και ξεπεράσει την πάρα του 3%. Η Ουγγαρία ισχυρίζεται ότι μετά το 2012-2013 το έλλειμμα δεν θα ξεπεράσει το 3%. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά. Όταν βλέπουμε όλα αυτά τα νέα μέτρα, την ρεσιμότητα, τα μακροοικονομικά κριτήρια, όλα αυτά τα νέα κριτήρια, Πρέπει να δούμε σε ποιο βαθμό οι κυρώσεις είναι βάσιμες, έχουν νόημα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την περίοδο μετά το 2014. Αλλά εδώ υπάρχουν προβλήματα. Βασιζόμαστε στην απόφαση που πήρε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρυσι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίρνει αποφάσεις που σκοπό έχουν να τιμωρήσουν μια χώρα. Και νομίζω ότι βασίζεται σε δεδομένα που δεν είναι αξιόπιστα. Μην ξεχνάμε ότι εδώ παίζεται όλο το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Μην ξεχνάμε ότι η απόφαση της Επιτροπής λέει ότι η πολιτική συνοχής δεν είναι ένα μέσο ανάπτυξης, αλλά είναι μια βοήθεια, μια επιδότηση. και οι επιδοτήσεις αυτές θα ανασταλούν. Το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό. Νομίζω ότι τους επόμενους μήνες θα πρέπει να αναλύσουμε την απόφαση που έλαβε την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί δημιουργείται ένα προηγούμενο. Μπορεί δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί στο μέλλον να χρησιμοποιεί κατ' επανάληψη αυτό το όπλο και μάλιστα χωρίς να βασίζεται σε αξιόπιστα στοιχεία. Αυτό μας ανησυχεί. Είναι μια απόφαση η οποία δεν είναι σωστή αυτή η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κ. Φασάκας θέλει να αντιδράσει και να παρεύει και αυτό στη συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Ντανούτα. Εξάρτητα πόσο χρόνο έχετε. Με μεγάλη χαρά να αντιδράσω κι εγώ. Θέλω να σε ευχαριστήσω εσάς και όλα τα μέλη της, ε, Ευρωπα... της ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που εκτιμάτε την ε, γνωμοδότησή μας. Είναι πολύ σημαντικό να αλληλοϊποστηριζόμεθα, αλλά πριν την αλληλοϊποστήριξη πρέπει να σας πω ποια είναι η θέση μας. Εσείς είσαστε πολιτικοί, παίρνετε πολιτικές και νομοθετικές αποφάσει. Εμεί διαμορφώνουμε κάποιες γνώμε. Η οι γνώμες μας δεν είναι πολιτικού χαρακτήρα, αλλά έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα. Και αμφισβητούμε τις αποφάσεις. Ελπίζουμε λοιπόν, υπ' αυτή την έννοια, η γνωμοδότησή μας να σας υποστηρίξει. Ελπίζουμε όλα αυτά να τα λάβετε υπόψη σας, ούτως ώστε να τα εντάξετε στον τελικό κανονισμό. Μόνο έτσι μπορεί να σας βοηθήσει το ελεκτικό συνέδριο. Με μεγάλη χαρά λοιπόν είδα ότι οι περισσότεροι από εσά για το ανώτατο όριο, για τις μακροοικονομικές ε, προϋποθέσεις, για τις μειώσεις κτλ. Ε, κινούμαστε προς την ίδια κατεύθυνση. Και νομίζω ότι το ίδιο θα ισχύσει και με την ε, Επιτροπή Κοκομπού. Όταν συζητήσετε με τις άλλες επιτροπές, μια και είσαστε η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή, μπορείτε να το πείτε αυτό ότι είμαστε στο ίδιο μήκο κύματο. Σε ό,τι αφορά το ανώτατο όριο, το ανώτατο ποσοστό, ε, λυπάμαι που ο Βίκτορ δεν ήταν εδώ, αλλά τον άκουσα με μεγάλη προσοχή και νομίζω ότι ανέφερε ακριβώ τα ίδια που, μιλάμε, που λέμε και εμεί για τη μείωση του ανώτατου ορίου. Αν η Κομισιόν λέει, το οποίο δεν είναι σωστό, ότι λόγω του 4% που προβλεπόταν για αυτή την περίοδο, ε, επειδή δεν μπορούσε να απορροφηθεί αυτό, τώρα κάνουμε μια γενική μείωση. Κοιτάξτε, σας παρακαλώ, πέστε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πριν προβείτε σε τέτοιες ε, μειώσει, πέστε μα ποιοι είναι οι λόγοι. Είναι περιορισμοί στον προπολογισμό, υπάρχουν άλλα προβλήματα. Τα, τα χρήματα δεν υπάρχουν για να τα αποταμιεύουμε, αλλά να τα ξοδεύουμε για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και για τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Το άλλο που είπε ο Βίκτορ, αν, αν το μειώσουμε στο 2,5% θα υπάρξει τεράστια διαφορά ανάμεσα στις στοχές και στις ε, πλούσιες χώρες. Ο βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής είναι να βοηθήσουμε τις στοχές χώρες να αποκτήσουν περισσότερες ευκαιρίες με ευρωπαϊκά κονδύλια, με τα χρήματα της πολιτικής συνοχής να αναπτυχθούν. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η μείωση θα πρέπει να εξεταστεί περισσότερο. Είπατε ότι δεν είστε συνηθισμένοι να μιλάμε τόσο ανοιχτά εμείς ως ελεγκτικό συνέδριο. Κοιτάξτε, Έχουμε τις νομοδοτήσεις, τις γραπτές. Αυτό είναι μια απόφαση της 16ης-15ης ε, Δεκεμβρίου. Είναι η γνωμοδότηση του ελεγκτικού συνεδρίου. Κατά τύχη εγώ είμαι Ούγγρος και την παρουσιάζω. Αλλά αυτή είναι η γνωμοδότηση του ελεγκτικού συνεδρίου που ε, υιοθετήθηκε ομόφωνα από το σώμα των μελών του ελεγκτικού συνεδρίου. Τώρα ας πάμε στις ε, μακροοικονομικές προϋποθέσεις. Κρίσιμο θέμα. Ως ελεγκτικό συνέδριο είπαμε ότι το six-pack είναι ένα σύστημα όπου οι μακροοικονομικές προϋποθέσεις συζητώνται μαζί με τις χώρες. Αν και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει περίπτωση η χώρα να χρειαστεί να πληρώσει ένα πρόστιμο. Ξέρετε πολύ καλά επίσης ότι συζητάμε με τους δικαιούχους σε περίπτωση που σταματάμε την ε, καταβολή της πληρωμής. Αν η χώρα έχει ε, τεράστια προβλήματα, έχει προβλήματα με τις επενδύσεις, με τα προγράμματα, με τις ε, περιφέρειες, Τι γίνεται τώρα, τότε. Θα αναγκάσουμε τη χώρα να πληρώσει, γιατί τα project είναι εν εξελίξη και σε αυτήν την περίπτωση το έλλειμμα όμως θα αυξηθεί ή θα πρέπει να σταματήσετε τα προγράμματα, τα project. Αλλά τότε υπάρχει τεράστια ασφάλεια νομική, τεράστια ασφάλεια δικαίου. Γιατί οι συμβάσει έχουν υπογραφεί. Ποιο κάποιο πρέπει να πληρώσει. Γι' αυτό λοιπόν μα είπε το ελεκτικό συνέδριο. Προσοχή, προσοχή. Δεν είναι το σωστό μέτρο αυτό. Δεν πρέπει να τα μπερδεύετε ε, αυτά. Γιατί έτσι ξεχνάτε ποιος είναι ο βασικός στόχος της ε, πολιτικής συνοχής. Σε αυτά που είπε ο εισηγητής, περιμένω τη συζήτηση την Τετάρτη στην Κοκομπού, στην Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών και ελπίζω για τα ειδικά θέματα να φτάσουμε σε μια κοινή θέση, σε ενιαία συμπεράσματα και ελπίζω αυτό να σας βοηθήσει και εσάς για να υιοθετηθεί το συντομότερο δυνατό ο τελικός κανονισμός. Νίκολας Μάρτ. Ο Νίκολας Μάρτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μου δίνετε την ευκαιρία να πω δύο λόγια ως απάντηση στις παρατηρήσεις του κ. Φαζάκας. Καταρχήν, αντιλαμβάνουμε πως η ανάλυση της νομοδότησης του Ελληνικού Συνεδρίου είναι πολύ προσεκτική και πολύ αντικειμενική στην αξιολόγηση του πακέτου για τα ταμεία. Η γνωμοδότηση του Ελληνικού Συνεδρίου αναφέρει βέβαια πολλά θετικά πράγματα, κάτι που δείχνει ότι η Κομισιόν έχει κινηθεί προ την ορθή κατεύθυνση. Όπω είπε ο κ. βέβαια σήμερα δεν έχουμε πολύ χρόνο για να μπούμε στι λεπτομέρειε. Είναι πολύ χρήσιμε οι παρατηρήσει ε, του Ελεκτικού Συνεδρίου. Τις έχουμε λάβει υπόψη, τις σκεφτήκαμε ήδη και σίγουρα θα σα εξηγήσουμε ποια είναι τα συμπεράσματά μας, αλλά να εστιατώ σε αυτά τα τέσσερα θέματα που οποία Πρώτον, για το θέμα της ευρωπαϊκής προσθέμενης αξίας και την εστίαση στα αποτελέσματα. Δεν έχουμε μετακινηθεί πλήρως σε ένα τέτοιο σύστημα, το εξετάζουμε ε, δεν πιστεύουμε ότι θα λειτουργήσει για την πολιτική συνοχή να μετακινηθούμε σε ένα σύστημα που θα είναι ε, καθαρά εστιασμένο στα αποτελέσματα. Βέβαια, προτείνουμε κάτι που μετακινείται από την σημερινή προσέγγιση των input προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν υπόψη μια καινούργια λογική παρέμβασης. Αυτό δεν είναι μονολόγια, έχει ε, ενταχθεί στο μηχανισμό στρατηγικού σχεδιασμού και με αυτόν τον ε, τρόπο μπορούμε να αναστείλουμε πληρωμές και να επιβάλλουμε διορθώσεις όταν οι στόχοι δεν πληρούνται. Έχουμε λοιπόν τα μέσα που χρειαζόμαστε και ένα σύστημα κινήτρων που θα ενισχύσει την παρακολούθηση. Συνεπώς, νομίζω ότι έχουμε μια δομή ήδη ετοιμάσει που αντικατοπτρίζει μια τελείω διαφορετική προσέγγιση πια. Σε ό,τι αφορά την αριθμότητα εξάντεκτων των προτέρων, καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα αποτελούσε μια τέτοια αριθμότητα θα αποτελούσε σημαντική αλλαγή και θα μας βοηθούσε στο να δημιουργήσουμε την κατάλληλη βάση για τα αποτέλεσματα που θέλουμε. Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των κατεξιοδότηση και των κατεφαρμογή πράξεων, ε, δεχόμαστε ότι θα πρέπει να δικαιολογούμε κάθε φορά τις ε, επιλογές που κάνουμε, όπως και στο παρελθόν ορισμένα τεχνικά στοιχεία θα πρέπει να ρυθμίζονται σε ένα δεύτερο επίπεδο πράξεων, αλλά νομίζουμε ότι η πρόταση της ε, Κομισιόν έχει πετύχει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στις ε, επιθυμίες του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει βέβαια να εξασφαλίσουμε ότι η κατεξοδότηση πράξης θα είναι λογικά συνεπής και θα παρουσιάσουμε τα βασικά στοιχεία μας, θα παρουσιάζουμε τα βασικά στοιχεία κάθε ε, τέτοιας πράξης. Σε ό,τι αφορά το το ανώτατο όριο και την μακροοικονομική ρεσιμότητα. Ε, το ανώτατο όριο, η οροφή, αποτελεί τμήμα μια συνολική αξιολόγηση τη ε, ε, Κομισιόν στο πλαίσιο του πολιτικού δημοσιονομικού προγράμματος ε, προκειμένου να ε, είμαστε σίγουροι ότι ε, θα εξασφαλίσουμε μια συνολική ισορροπία. Συνεπώ, η οροφή δεν θα πρέπει να ειδωθεί αποκομμένα, αλλά στο πλαίσιο Τη συνολική πρότασης τη Κομισιόν. Ένα στοιχείο ήταν η απορροφητικότητα. Δεν ήταν το μόνο στοιχείο. Άλλωστε η Κομισιόν έχει υπόψη της ότι ακόμα και η, ε, τα διαφοροποιημένα ποσοστά ε, απορρόφησης ε, μπορούν επίσης να κατακριθούν και έχουν αντεπιχειρήματα. Νομίζω ότι η ανώτατη ροφή είναι δικαιολογημένη συνολικά, βέβαια Σίγουρα θα πρέπει να το εξετάσουμε και να το υποστηρίξουμε από τη δική μα πλευρά στι διαπραγματεύσει για το δημοσιονομικό πλαίσιο. Σε ό,τι αφορά τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα, επιμένουμε σε αυτή την πρότασή μας, θα την υποστηρίξουμε και για να χρησιμοποιήσω την αναλογία του κ. Φαζάκας, δεν έχει σχέση με την ε, ε, αφαίρεση ε, του φαρμάκου που ένα άρρωστο ασθενή. Όχι. Η, η αρχική ε, κατάσταση είναι ένας ασθενής ο οποίος δεν παίρνει το φάρμακο που του δίνουμε. Γιατί πάντοτε ξεκινάμε αυτή τη διαδικασία για κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν συμμορφωθεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις. Και πάντοτε είναι μια απόφαση του Συμβουλίου αυτή που ξεκινάει οποιαδήποτε δράση ε, αναστολής ε, δεσμεύσεων και πληρωμών. Δεύτερον, ε, ε, αναφέρθηκε μια πρόσφατη απόφαση για την διακριτική ευχέρεια που υπάρχει για να εξασφαλίσουμε την αναλογία, την αναλογικότητα, συγγνώμη, και για το ότι είναι δυνατόν η εφαρμογή να γίνει εστιασμένα έτσι ώστε να μην προκύψουν Ε, ανεξέλεγκτες ε, συνέπειες ε, για αυτούς που είναι καλά προετοιμασμένοι και υλοποιούν σωστά τα προγράμματά τους. Οπότε, αν δούμε την αναστολή των δεσμεύσεων, των μισθώσεων δεσμεύσεων, στην Ουγγαρία, το αποτέλεσμα, καταρχήν, θα φανεί το επόμενο έτος από αυτό το δεσμεύσεων, δηλαδή το 2013. Αλλά ακόμα και τότε δεν θα είναι άμεσο, άμεσο ο αντίκτυπο, το αποτέλεσμα, διότι θα γίνει σαφής ο αντίκτυπος μόνον αφού εξαντληθούν οι πιστώσεις δεσμεύσεων. Τότε μόνο θα έχει δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Συνεπώ, θα περάσει αρκετό χρόνο και κατά τη διάρκεια αυτή τη περίοδου το κράτο μέλο μπορεί να αναλάβει τη δράση έτσι ώστε ε, να εξασφαλίσει την άρση αυτή τη αναστολή. Επίσης να σας πω ότι αυτό είναι μια πρόταση της Κομισιόν, δεν είναι μια απόφαση. Η απόφαση θα ληφθεί από το Συμβούλιο τελικά. Ευχαριστώ. Σα ε, Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Φυσικά το θέμα μακροοικονομικής ρεσιμότητας δεν έχει να κάνει μόνο με δεσμεύσεις, αλλά και με πληρωμές. Είναι λοιπόν πιο δύσκολο. Και έτσι θα ήθελα να κλείσω και το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη και να περάσω γρήγορα γρήγορα σε αυτό που ήδη ξεκινήσαμε, τη συζήτηση για κάποια θέματα του γενικού κανονισμού να, ζητήσω το, να δώσω το λόγο κατευθείαν στο Λαμπέρ και να θέσει τα ζητήματα που τα αγαπάει πιο πολύ από όλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω καταρχάς ότι η κυρία Κρέλ δεν είναι εδώ σήμερα γιατί είναι άρρωστη. Θέλει να έρθει εδώ πέρα στη συζήτηση, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί σήμερα. Δεν ξέρω, είναι το σύνδρομο με τι απόκριε. Δεν ξέρω τι είναι. Τέλο πάντων, ελπίζω να τα πάει καλά, να αναρρώσει γρήγορα τώρα σε πιο σοβαρό επίπεδο. Έχουμε την ευκαιρία να εξετάσουμε διάφορα σημεία ε, που έχουμε ήδη εξετάσει στο παρελθόν. Από τα 11 σημεία έχουμε ε, ήδη εξετάσει εκ το και έχουμε λοιπόν κάποια που απομένουν και μετά μπορούμε να περάσουμε στη διαδικασία την υπόλοιπη. Κατάρχά η διαδικασία είναι η εξή. Είμαστε επιτεθειμένοι να εργαστούμε στο χρονοδιάγραμμα, στο οποίο σας έχουμε ήδη διαβιβάσει. Να σας υπενθυμίσω ότι τώρα εξετάζουμε το έγγραφο, αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να το εξετάζουμε. Πρέπει να προβούμε σε κατάθεση της έκθεσης τροπολογίας. 20 Μαρτίου λοιπόν έχουμε την ακρόαση. Αυτή είναι σημαντική ημερομηνία γιατί λαμβάνουμε υπόψη διάφορες μελέτες και διάφορα άλλα σημαντικά στοιχεία και είναι ανοιχτό για όλους αυτό το, αυτή η εκδήλωση. Μετά έχουμε το σχέδιο έκθεσης. Στα αγγλικά θα το έχουμε ήδη στις 26 Απριλίου ή στις 8 Μαΐου σε έκτακτη συνεδρίαση. Πρέπει να βιαστούμε. Το ακούσατε και πριν από λίγο ότι από πλευρά περιεχομένου θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Γιατί άλλο θα χάσουμε. Προθεσμία για την καταθέση τροπολογιών το Μάιο, θα πρέπει να βεβαιωθεί και αργότερα αυτό, και μετά εξέταση των τροπολογιών τον Ιούνιο και η έγκριση στην Επιτροπή Ρέτζη 11 Ιουλίου. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν εργαζόμαστε. Φυσικά έχουμε κάποιες ευκαιρίες για συζήτηση. Να τονίσω το σημείο 11 καταρχάς. Η σύνδεση της, ε, του Europe Facility Έχουμε συζητήσει πώς σχετίζονται όλα αυτά με την κοινή διαχείριση, γιατί πάντα μιλάμε υπό το πρίσμα της συνοχής. Πώς μπορούμε λοιπόν να βάλουμε μια κεντρική αρχή να τα διαχειριστεί αυτά. Γιατί δεν είναι σαφές πώς θα επιστρέψουν οι πόροι. Είναι σαφές ότι τα χρήματα ότι οι πόροι επιστρέφουν στις χώρες συνοχής, αλλά πώς μπορούμε να τα αφαιρέσουμε από τους στόχους τους οποίους έχουν ανατεθεί. Φυσικά θα πρέπει να κοιτάξουμε θέματα ποιότητας. Δεν είναι όμως δίκαιος τρόπος αυτός απαραίτητα να απορροφούν μια-δυο χώρε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των ποσών αυτών. Αυτό θα το συζητήσουμε. Όπως και να έχει, η κυρία Κρέλ και εγώ αποδεχόμαστε το γεγονός ότι μεταφέρεται σε αυτό το connectivity facility. Έτσι έχει η κατάσταση λοιπόν σήμερα. Κάτι άλλο πιο τεχνικό που συζητάμε και σε ό,τι αφορά το κάπινγκ, τα ανώτατα όρια. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί ξέρετε, όταν αφαιρούνται οι πόροι, πώς επηρεάζει αυτό τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Αυτή λοιπόν είναι η θέση μας. Εντάχει, επί του παρόντος, ε, το αποθεματικό απόδοσης θα διατηρηθεί. Μάλλον αυτό θα εμείνουμε στην θέση μας, που είναι επικριτική. Δεν θεωρούμε ότι αν υπάρχουν τόσο μεγάλα προβλήματα, αν υπάρχουν οι όροι εξάντε, αν έχουμε συμφωνήσει επί των κριτηρίων απόδοσης για κάθε χώρα, αν υπάρχουν συμφωνίες εταιρικές, εταιρικής σχέσης, όπου η επιλογή χωρών συνάδει με αυτά που έχουν αποφασιστεί, γιατί χρειαζόμαστε, για ποιο λόγο χρειαζόμαστε αποθεματικό ε, απόδοσης. Ε, Αιδίες. Δεν θεωρώ ότι μας ε, αποφέρει το οτιδήποτε παρά θέμενη γραφειοκρατία. Γραφειοκρατία. Τίποτα παραπάνω. Δεν συμφωνούμε. Εμάς μας αρέσει πιο πολύ αυτά που προτείνει η Επιτροπή των Περιφερειών. Να πούμε ότι αν υπάρχουν πόροι που δεν έχουν δαπανηθεί, αυτόματα αποχαρακτηρίζονται και χρησιμοποιούνται για άλλα project εντός, εντός της χώρας. Ε, ίσως αυτό λοιπόν αποτελεί πιο αποτελεσματική λύση παρά το να πιέζουμε για ένα αποθεματικό απόδοσης. Δεν είναι πάντα ο καλύτερος μαθητής στην τάξη αυτό αυτό τον οποίο θα πρέπει να δώσουμε την πιο πολύ προσοχή. Αυτό λέει πάντα στα παιδιά μου. Κάτι άλλο που αναφέραμε σήμερα για τα ανώτατα όρια, για το κάπινγκ. Η αίσθησή μου είναι μετά από αυτά που ακούσαμε Αυτό θα συζητηθεί στο πολυετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο και στη σχετική επιτροπή στο Συμβούλιο. Εμείς θα πρέπει να παρουσιάσουμε την δική μας άποψη. Δεν νομίζω όμως ότι μπορούμε να λάβουμε την τελική απόφαση. γιατί αυτό ίσως να είναι αντιπαραγωγικό σε κάποιες περιπτώσεις σε σχέση με τους στόχους της Ευρώπης. Θα πρέπει να γίνει μια τελική συζήτηση για ένα πιο ισορροπημένο αποτέλεσμα από αυτό που έχουμε σήμερα. Γιατί για κάποιες χώρες υπάρχουν κάποια μη ηθελημένα αποτελέσματα που δεν παρέχουν ισορροπία τώρα κατά πόσον μπορούμε να το λύσουμε εμείς αυτό μέσω πρώτης ανάγνωσης δεν ξέρω. Ίσως θα μπορούσαμε να επιλύσουμε ένα 90% των υποθέσεων. Και τέλος, ε, πρόεδρε, ο Γιάνν Όλμπρεχτ από το Περιφερειακό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης δεν είναι εδώ σήμερα και ζήτησε τα τεχνικά αυτά ζητήματα, τα νέα αυτά εργαλεία στην αστική διάσταση να συζητηθούν μαζί του. Έχω την αίσθηση ότι με την ακρόαση μπορούμε να προβούμε σε κατάθεση τροπολογιών. Αν υπάρχει κάτι ωστόσο που δεν το έχουμε προσέξει και εγώ και η κυρία Κρέλ, να μας το επισημάνετε για να είμαστε καλά προετοιμασμένοι. Ο κύριος Γκουτμάνης. Το μικροφόνο. Ε, regarding performance reserve. Σε ό,τι αφορά το αποθεματικό απόδοσης. Μέχρι τώρα έχουμε 5% μέχρι το τέλος της περίοδου αν η χώρα ε, δεν έχει παρουσιάσει ατασταλίες, θα πάρει και το 5% του τελευταίο. Αν όχι, δεν το λαμβάνει αυτό. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι γίνεται με το 5% αυτό στο μέσο της περίοδου από μαθηματικής, από μαθηματικής άποψης. Ποιο θα είναι το κριτήριο αν δεν, τα έχει, αν δεν έχει πετύχει η χώρα. Κοιτώντας τα πραγματικά ποσά, υπάρχει μεγάλη ε, ε, διαφορά μεταξύ χωρών, μέχρι το 300% σε ό,τι αφορά την απορροφησιμότητα. Αλλά νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμένει στο παθηματικό αυτό, ενώ το βασικό ερώτημα είναι ποια θα πρέπει να είναι τα κριτήρια που θα πρέπει να οριστούν πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, γιατί αν αλλάξουν τα κριτήρια αυτά κατά τη φάση της εφαρμογής, της υλοποίησης, τα αποτελέσματα θα είναι οδυνηρά. Και εδώ θα συμφωνήσω με τον εισηγητή. Τι είναι χειρότερο, τα κριτήρια απόδοσης να οριστούν από το τέλος μέχρι το μέσο, μέσω της προγραμματικής περίοδου. Είμαστε πολύ φιλελεύθεροι ωστόσο, γιατί όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει την περίοδο 2000-2006, γιατί υπάρχουν κάποιες χώρες που ακόμα και σήμερα δεν έχουν, τους έχει αφαιρεθεί το 5%, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιμένει να ολοκληρωθεί πλήρως η φάση της εφαρμογής για το Connection Facility. Το ερώτημα είναι γιατί συνδέεται η πολιτική συνοχή με τα δύο αυτά ζητήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να φρεθούν 10 εκατομμύρια από την, δισεκατομμύρια από την ε, πολιτική συνοχή. Το θέμα είναι λοιπόν γιατί έγινε αυτή η πρόταση. Δεν νομίζω ότι έχουμε ιδιαίτερα επιχειρήματα κατά της πρότασης, αλλά το θέμα είναι πώς θα λειτουργήσει η κοινή διαχείριση. Γιατί είναι πολύ διαφορετική η διαχείριση των προγραμμάτων σε σχέση με τα προγράμματα συνοχής που έχουμε εδώ. Για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. το που είπε στο τέλος ο κύριος Φανίστελτρο για το κάπινγκ, για τον ορισμό των ανώτατων ορίων. Και εγώ έχω εργαστεί στο Συμβούλιο σε κάποιες περιστάσεις. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι το εξή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχει ομοφωνίες. Κάποιες χώρες θα είναι υπέρ, κάποιες θα είναι κατά. Από ρεολεστική άποψη η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι αυτή που θα αποτελέσει τη βάση του συμβιβασμού. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι βάσει τη πρόταση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να εργαστούμε. Δεν φαντάζομαι να υπάρχουν τεράστιες αλλαγές, ούτε ε, αυξητικέ ούτε μειωτικέ. Αλλά αν κανείς δεν μπορούσε να συμφωνήσει με τους άλλους, ε, σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει συμφωνία, η πρόταση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είναι το ουδέτερο έδαφο αν θέλετε. Και τέλος, μιλώντας για το τι συμβαίνει σήμερα. Σήμερα τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά, κυρίες και κύριοι. Όλοι είδαμε τα θετικά αυτά στοιχεία για το πώς θα έχουν ολοκληρωθεί οι πληρωμές μέχρι το τέλος του 2011 και σε πληρωμές και σε δεσμεύσεις. Αλλά από φέτος έχουμε μεγάλα προβλήματα γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει έλλειμμα και το έλλειμμα στις αρχές του έτους ήταν 15 δισεκατομμύρια περίπου. Τώρα έχει μειωθεί κάπως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι θα είναι πιο περιορισμένα, αλλά και πάλι είναι τεράστιο το ποσό. Πώς θα καλυφθεί αυτό το έλλειμμα λοιπόν. Να μην αναφέρω χώρες που δεν, που δεν έχουν πληροφορίες, αλλά κάποιες χώρες έχουν διακοπή, αν θέλετε, ε, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Όχι επειδή υπάρχει πρόβλημα, αλλά επειδή υπάρχει έλλειψη πόρων από πλευρά τη Επιτροπή. Εγώ θεωρώ ότι ο μοναδικό τρόπο ε, βελτι... Ε, ρύθμιση και διόρθωσης του προβλήματος είναι με την τροποποίηση των προπολογισμών. Η κατάσταση όμως είναι πάρα πολύ σοβαρή και για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Γιατί αν βρεθούμε σε μια κατάσταση που δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι, δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι χρηματοδοτήσεις, μιλάμε για δέκα δισεκατομμύρια έλλειμμα και δεν έχουμε και πάρα πολλού πόρους. Έχουμε, στο παρελθόν είχαμε δύο πηγές από προγράμματα που δεν πραγματοποιήθηκαν, αρωτικά προγράμματα που δεν ε, πραγματοποιήθηκαν και από την ανάπτυξη. Και τώρα, στο τέλος του δημοσιονομικού πλαισίου, όλοι θέλουν να ανακτήσουν αυτούς τους πόρους δεδομένου του ελλείμματος. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Νομίζω ότι καλύτερα είναι να αλλάξουν οι προϋπολογισμοί για το τρέχον και το επόμενο έτος, γιατί ιδάλλως, εξ όσων γνωρίζω, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινήσει να κοιτάει καταρχάς Πρώτο παράδειγμα, των, τις, ε, αρχές κοινού ελέγχου στα κράτη-μέλη. Δυστυχώς δεν αναπτύχθηκαν 100% ε, κοινέ τέτοιες αρχές ελέγχου. Υπήρχαν τέτοιες προθέσεις, αλλά αυτό μετατίθεται ως πρόβλημα στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Ιδάλλως ε, μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίσει ότι δεν είναι καλός ο κοινός έλεγχος γιατί δεν υπάρχει σχετικές, ε, δεν έχουν οριστεί σχετικές αρχές. Κατά δεύτερο, το θέμα των συστημάτων ελέγχου διαχείρισης. Αν πιστοποιείται ένα σύστημα ελέγχου προγραμμάτων, σημαίνει αυτό τι, ότι το έχει αποδεχτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν κατά τη φάση της εφαρμογής, λόγω έλλειψης κονδυλίων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινήσει να λέει ότι, «Αν κοιτάξτε, θα πρέπει κάτι να αλλάξετε στο στο MSC e». Αυτό είναι προβληματικό. Το θέμα είναι αυτές οι πρακτικές να μην μεταφερθούν στις επόμενες δημοσιονομικό πλαίσιο και στη τελική ανάλυση η πρότασή μου είναι η εξή. Δεν πιστεύω ότι είναι θέμα ούτε ελέγχου, ούτε συστήματος ελέγχου και κατά δεύτερον, αν το σύστημα ε, διαχείρισης έχει οριστεί, έχει οριστεί γιατί κάποιες χώρες έχουν ε, κάποια αποκεντρωμένες υπηρεσίες, άλλες έχουν κάποιο υπουργείο. Όλα αυτά δεν μπορούν να αλλάξουν στη φάση της εφαρμογής και μιλάμε ναι, ναι, για την επόμενη περίοδο. Αυτό προτείνω προς τον εισηγητή. Ευχαριστώ. One more speaker, Τελευταίος ε, εισηγητής και αύριο θα συνεχίσουμε ε, να συζητάμε αυτή την έκθεση μετά τις ψηφοφορίες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ως ε, σκιώδης εισηγήτρια για το Γεωργικό Ταμείο και για, τους, και για το Connecting Europe Facility. Θέλω να μιλήσω για τα άρθρα 14 ε, και 84 του Γενικού Κανονισμού. Άρθρο 14 καταρχάς. Ε, οι συμβάσεις εταιρικής σχέσης. Έχουμε μία... Θέλω να ρωτήσω μάλλον ποια είναι η προστιθέμενη ε, αξία από τη δημιουργία μιας πλατφόρμας εάν ε, συνεχιστούν οι ανταλλαγές όπως το Ιρμπάκ. Ε, όταν δεν έχουμε ε, ολοκληρωμένη στρατηγική για τις πόλεις. Τι σχέση έχει αυτή η πλατφόρμα με τις καινοτόμες αξίες ε, στα πλαίσια του Ουρμπάκ που δεν υποφελούνται από την ολοκληρωμένη στρατηγική ή στρατηγικές. Σε αυτό το άρθρο η Κομισιόν προτείνει τη δημιουργία εδαφικών επενδύσεων που ε, υπέρ των πόλεων υποτίθεται. Εγώ φοβάμαι ότι αυτό το νέο εργαλείο ε, περιπλέκει την σχέση τα, μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων. Αν η Κομισιόν δεν ζητήσει περισσότερες επιδοτήσεις γενικά αυτό το εργαλείο θα είναι επιζήμιο. Μιλάμε τώρα για τα κέντρα των πόλεων, για δύσκολες περιοχές. Για το άρθρο 84. Πώς ε, έφτασε η Κομισιόν σε αυτά τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Συνοχής. Ίσως υπάρχει, εδώ υπάρχει τεράστιο πρόβλημα ε, διαφάνειας. Υπάρχει έλλειψη διαφάνειας και για το νούμερο και για τον ορισμό των αξώνων προτεραιότητας, ειδικά σε ό,τι αφορά τις μεταφορές. Υπάρχει τεράστιος κίνδυνος. Νομίζω ότι η πολιτική, το λέμε και το ξαναλέμε, υποτίθεται ότι γίνεται από κάτω προς τα πάνω. Εδώ όμως δεν εξασφαλίζεται αυτό το αυτή η επίπεδη διαχείριση. Επίσης, το 0,2% των πόρων του Γεωργικού Ταμείου υπέρ των καινοτόμων δράσεων για την ε, ανάπτυξη των πόλεων. Πώς ε, υπολογίσατε τις ανάγκες αυτές των πόλεων, ποιες είναι οι εγγυήσεις για τα προγράμματα που επιλέγονται, τα προγράμματα αυτά είναι μεγάλα προγράμματα ή όχι μόνο, χρειάζονται μεγάλη χρηματοδότηση ή όχι. Αυτά τα προγράμματα δεν θα πρέπει να προωθούν την έξυπνη ανάπτυξη. Δεν θα πρέπει να είναι υπέρ της καταπολέμησης της στόχιας, της κοινωνικής ένταξης. Υπάρχει και εδώ τεράστια έλλειψη διαφάνειας. Ε, κύριε Φανίλθεροι, έχετε πληροφορίες για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε εδώ, συνάδελφοι. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 9 και θα συζητήσουμε αυτό το σημείο μετά την ψηφοφορία. Ο κύριος Φανής Τελρόη, μία παρατήρηση, παρακαλώ. Πρόεδρε, δεν έχει να κάνει με το μήκο τη συζήτησή μα, το γεγονό ότι δεν ολοκληρώνουμε τώρα, να σα πω ότι αμέσω μετά την ψηφοφορία αύριο θα πρέπει να μεταβώ στην Επιτροπή Ήτρε για να ψηφίσω. Μήπω να το βάλουμε κάποια στιγμή την πρώτη ώρα για να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις για την αστική διάσταση. Είναι πολύ καλή αυτή η παρατήρηση. Γιατί εκεί ακριβώς ορίζεται τέτοια θέματα. Για να δούμε μήπως μπορούμε να το κοιτάξουμε 10 παρατέταρτο πήγε το θέμα, να δούμε ποιοι θέλουν να μιλήσουν. So we Ναι, θα το προσπαθήσουμε. Γεια σας. Δεν μπορούμε να είμαι παρόν αύριο. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον πάντως ε, όλα όσα υπόθηκαν για αυτό το σημείο και για τα υπόλοιπα σημεία, αλλά ξέρετε ότι η έδρα μας είναι στο Λουξεμβούργο και δεν μπορούμε να ξανάρθουμε. Πάντως θέλω να σας πω ότι μας αρέσει η πρότασή σας. Καλή τύχη. Ελπίζω να ενταχθούν όλα αυτά τα στοιχεία στην τελική έκθεση. Δυστυχώς βέβαια ε, η θέση σας δεν συμπεριπτεί πάντα με τις Κομισιόν. Ελπίζω να περάσει η δική σας θέση, η δική σας άποψη. Μην ξεχνάτε ότι θα σας χρειαστούμε και για τις επόμενες ε, διαδικασίες απαλλαγής, τα επόμενα χρόνια. Θα σας ξαναδούμε λοιπόν.